Καλημέρα λοιπόν. Σας, ε, σας χαιρετίζω στην τελευταία, μάλλον στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού. Αν δεν έχετε καμία αντίρρηση μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Έγκριση των πρακτικών 15-16 Ιουνίου. Εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του πακέτου για την Ενεργειακή Ένωση, στρατηγική πλαίσιο και πρωτόκολλο των Παρισίων με την κυρία Βίρκουνεν και τον κύριο Έικχαουτ, οι οποίοι είναι συγητές και τους δίνω το λόγο καταρχήν στην κυρία Βίρκουνεν. Έχετε το λόγο λοιπόν. ευχαριστώ και... Ε, ευχαριστούμε και όλους τους σκιώδες ηγητές και όλα τα μέλη της Επιτροπής των Μεταφορών. Έχουμε 56 τροπολογίες, 7 συμβαστικές τροπολογίες. Γιατί συνοηθήκαμε πάρα πολύ καλά με τις πολιτικές ομάδες και τους κοιόδες ηγητές. Τους ευχαριστώ όλους για τη συμβολή τους. Και ακριβώς όπως συζητούσαμε προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς ως Επιτροπή να επικεντρωθούμε στα θέματα μεταφορών. Γιατί είναι δική μας αυτή η γνωμοδότηση και όπως γνωρίζετε στο σχεδίο κειμένου δεν αναφέρονταν τίποτα για τις ε, μεταφορές οπότε και είπαμε σε αυτές τις συμβαστικέ τροπολογίες εκεί να επικεντρωθούμε μόνο στα θέματα μεταφορών για τον ενεργειακό τομέα. Οπότε καλύπτονται σε αυτές τις συμβαστικέ τροπολογίες όλες οι τροπολογίες. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ όλους όσοι συνεργαστήκατε. Και ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα επιψηφίσει αυτές τις τροπολογίες. Πρόεδρος. Πολύ γρήγορα ήταν αυτά. Ο δεύτερος ηγητής όμως δεν είναι εδώ παρόν. Οπότε θα ζητήσω από τους κοιόδης να λάβουν το λόγο για το πρώτο αυτό η κυρία Γκρίφιν η πρώτη ούτε και η κυρία Γκρίφιν δεν είναι εδώ εδώ, ναι εδώ είμαι ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της νομίζω ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση η οποία θα δώσει ελπίζω προσθέμενη αξία στην τελική έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ Χάνα. Το ενεργειακό πακέτο είναι ένα σημαντικό νομοθέτημα το οποίο θα διαμορφώσει το στερέωμα ενεργείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση, στην ε, ανταγωνιστικότητα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη υπό την έποψη των μεταφορών. Οι μεταφορέ είναι ένα από του σημαντικότερου τελικού καταναλωτέ ε, ενέργεια και 94% των μεταφορών βασίζεται σε προϊόντα πετρελαίου. Εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα το όραμα τη Κομισιόν να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακο και πιστεύω ότι οι συγητές έχουν τονίσει σωστά την ανάγκη να προωθήσουμε την ηλεκτροκίνηση και την χρήση ηλεκτρισμού για να μειωθούν οι εκπομπές. Η αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας και η πρόθεση των ανανεωσίμων ενεργειών είναι πάρα πολύ σημαντική αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια πραγματική ενεργειακή μετάβαση. Για όλους αυτούς τους λόγους υποστηρίζω απόλυτα το να συμπεριλάβουμε δεσμευτικούς στόχους για την ενεργειακή απόδοση και την χρήση ανανεώσιμων ε, ενεργειών. Πιστεύω ότι αυτή η μετάβαση στα ενεργειακά θέματα θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο αν συμπεριλάβουμε και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το σύστημα διακυβέρνησης Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να είναι και εκ των κάτω προς τα άνω και εκ των άνω προς τα κάτω. Οι πολίτες θα πρέπει να βρισκόνται στον πυρήνα της Ενεργειακής Ένωσης. Είναι ευθύνη μας να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι οι ωφελημένοι από αυτή τη μετάβαση με το να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και με το να άρουμε τις ε, ανισότητες σε βάρος των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να περιλάβει και τις αστικές περιοχές και τις περιοχές της Υπέθρου. Χαίρομαι λοιπόν που η έχει καταθέσει μια πρόταση για να υποστηρίξει τη βιώσιμη κινητικότητα και σε επίπεδο αστικό και σε επίπεδο Υπέθρου για να μειωθούν οι πηγές ρήπανσης. Προσβλέπω λοιπόν στην άποψη όλων σας, αλλά και πάλι θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγητρία. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Ο Ιγνάσιο Φάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Βιρκούνεν και όλους τους συναδέλφους που ήταν σκιώδεις εισηγητές γιατί συνεργαστήκαμε με μεγάλη επιτυχία. 95% αφορά ε, προϊόντα ή υποπροϊόντα πετρελαίου. Οπότε αν θέλουμε κάτι να κάνουμε και αν θέλουμε να μην έχουμε διοξίδιο του άνθρακα ή άνθρακα στην οικονομία, τότε θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το ρόλο κλειδί των μεταφορών θα πρέπει να πούμε πώς θα έχουμε πιο αποτελεσματική μεταφορά της ενέργειας, τις μεταφορές, τι θα γίνει με το περιβάλλον, πιο καθαρές τεχνολογίες, το πώς υπάρχει διαλειτουργικότητα και άλλες τεχνολογίες, οπότε θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις πιο αποτελεσματικού τρόπους μεταφορών ε, για σιδηροδρόμους, για τους λιμένες και γενικά για τις συνδυασμένες πολυτροπικές μεταφορές, νότόμε τεχνολογίες, και επίσης να έχουμε κάποια έργα επίδειξης ε, κατά έναν ε, τρόπο που να καταλήγει ουδέτερο στην λογικό. Οπότε υπενθυμίζω σε όλους ότι η Ενεργειακή Ένωση είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ρόλο πρόκειται να παίξουν οι μεταφορές. Ελπίζω δε ότι αύριο θα έχουμε θετική ψήφο όλων των συναδέλφων και για άλλη μια φορά Ευχαριστώ την κυρία ε, Βίρκουνεν, την εισηγήτρια. Danke sehr. Jetzt Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Βίρκουνεν γιατί ήταν πάρα πολύ ε, επικοδομητική η συνεργασία μας ε, είχε πνεύμα συνεργασία, γι' αυτό κατέληξαν σε αυτού του συνδυασμού και τώρα όσον αφορά την Ενεργειακή Ένωση, πάνω σε αυτό θέλω και εγώ να σα μιλήσω, γιατί έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα. Θα πρέπει να δείξουμε την τόλμη να τα εξετάσουμε πρώτα-πρώτα. Το τι γίνεται με τα ορυκτά καύσιμα και πόσο τα στηρίζουμε δεν θα πρέπει να έχουμε διγλωσία. Γιατί από την άλλη μεριά θέλουν να προχωρήσουν και να μειώσουν τι πηγέ ενέργεια στην Ευρώπη. Οπότε να μην ε, προωθούμε τι παλιότερε τεχνολογίε, αλλά τι νεότερε. Αυτό να κάνουμε με την ε, ενεργειακή μας πολιτική. Θα πρέπει να έχουμε την ε, ενάργεια και να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σήμερα. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να θίξω είναι το εξή. Το δίκτυο διανομής για τους διάφορους ενεργειακούς πόρους. Είπαμε ότι αυτό είναι θέμα υποδομών στις μεταφορές. Θα πρέπει να περιχαρακώσουμε εκ νέου αυτή την πολιτική μας για να δούμε τι θα γίνει με το δίκτυο και πώς θα χρηματοδοτηθεί. θα πρέπει να είναι δημόσια χρηματοδότηση. Αλλά επίση θα πρέπει να κάνουμε κάτι και για ε, τις υπόλοιπες υποδομές. Φερρυπίν θα πρέπει να κατασκευάσουμε δρόμους. Οπότε και πάλι να ευχαριστήσω για την αγαστή μας συνεργασία. Ευχαριστώ κύριο Κλέζιτς. Ευχαριστώ κύριε Θα Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Βερικονέν καθώς και τους κοιότητες για τη συνεργασία. Ήδη έχουμε ακούσει πολλά για τη σημασία της ε, Ενεργειακής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα για τις μεταφορές στα πλαίσια της Ενεργειακής Ένωσης. Η ελεύθερη μετακίνηση είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να διαφυλαχθεί, να κατοχυρωθεί με βιώσιμο τρόπο βιώσιμες μεταφορές και άλλα θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών το ταχύτερο δυνατό, όχι μόνο για να μειώσουμε το έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ακριβώς των εισαγωγών ορεικτών καυσίμων αλλά και να συμβάλλουμε σε άλλους στόχους που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα παραδείγματος χάρη και προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που έχει αμεσοθετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Για τις ε, τροπολογίες, κάποιες δεν σταματώθηκαν στις συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ε, εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας ε, στην COP21. Ναι. Χρειάζεται Επίσης, να γίνουν επενδύσεις ανθρωπίνων πόρων και οικονομικών πόρων για την έρευνα, ούτως ώστε, όπως έλεγα, να ε, καταστούν βιώσιμες ε, οι μεταφορές ε, για τις σιδηροδρομικές και τις οδικές μεταφορές όλος ιδιαίτερες για να πρέπει να επιτύχουμε το ταχύτερο δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Πέρα από τις βιώσιμες μεταφορές υπάρχει ε, και μια βασική δραστηριότητα πολλών, ε, πολλών κρατών μελών, ο βιώσιμος τουρισμός και οι βιώσιμες ε, μεταφορές είναι βασική προϋπόθεση ώστε να είναι και βιώσιμος ο τουρισμός. Ελπίζω λοιπόν να υποστηρίξετε τη σχετική τροπολογία διότι Θα υποστηριχθούν έτσι όσοι έχουν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ στον τουρισμό. Ο Μπασάικο τώρα που ήρθε ο δεύτερος ηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που καθυστέρησα, γιατί είχα μια συζήτηση για την Ελλάδα. Κάτι φαίνεται να γίνεται εκεί. Αλλά έρχομαι στην COP21 στο Παρίσι. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε για το θέμα αυτό και θα ψηφίσουμε για αυτό το θέμα αύριο. Είναι χρήσιμο λοιπόν να ξέρουμε πού πηγαίνουμε με τις ε, τροπολογίες συμβιβασμού. Επτά τροπολογίες συμβιβασμού θα τεθούν επιτάπητος αύριο που καλύπτουν γενικά τις περισσότερες από τις τροπολογίες που προήλθαν από τις πολιτικές ομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους σκιώδεις για τις ε, επικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων ώστε να καταλήξουμε σε αυτές τις συμβαστικές λύσεις, τις οποίες οι περισσότερες πολιτικές ομάδες μπορούν να υποστηρίξουν. Δυστυχώς το EFDD και το ENF δεν ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και γι' αυτό δεν έχουν μάλλον δεν θα υποστηρίξουν τις τροπολογίες συμβασμού αλλά τα υπόλοιπα πέντε μεγάλα κόμματα υποστηρίζουν τις συμβαστικές λύσεις και χαίρομαι γιατί με τον τρόπο αυτό έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε μια συμφωνία. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας περισσότερο το θέμα των μεταφορών εν ώψη των διαπραγματεύσεων του Παρισιού. Ξέρουμε ότι το μέσο των μεταφορών επέχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο σοβαρά. Φυσικά δεν θα είναι στην κορυφή της ατζέντα το θέμα των μεταφορών, αλλά σίγουρα εμείς πρέπει να εστιάσουμε για τα θέματα μεταφορών και έχουμε λοιπόν μια μεγάλη παράγραφο για το ρόλο της ε, ΙΚΑΟ και του IMO, του Ναυτιλιακού Οργανισμού, που έχουν μεγάλο ρόλο και οι δύο φορέ για τη μείωση των εκπομπών και η συμβαστική λύση λέει ότι εμείς διαπιστώνουμε ότι επεξεργάζεται το θέμα αυτό, αλλά έχουμε ένα κριτικό πνεύμα σε σχέση με την έλλειψη πρόοδου που παρατηρείται στους οργανισμούς αυτούς. Αυτό είναι συμβαστική γλώσσα, δεν υπάρχει πιο συμβαστική. Τελικά όμως η δήλωσή μας είναι ότι η ΚΑΟ και ο IMO πρέπει να καταλήξουν σε κάτι το οποίο είναι θετικό, γιατί αυτοί οι τομείς της ναυτιλίας και της αεροπορίας θα πρέπει να συμβάλλουν <clears throat> σημαντικά για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο του να μην υπερβούμε τους δύο βαθμούς Κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας. Κατά τα άλλα έχουμε μια στεναρή διατύπωση και για το μέλλον των μεταφορών, για τους μηχανισμούς τιμολόγησης και την επίτευξη μιας ισορροπίας στο μείγμα ενέργειας που χρησιμοποιείται στον τομέα της ενέργειας. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν καλύπτονται από τις συμβαστικές λύσεις και θα δείτε στον κατάλογο ψηφοφορίας ότι αν ψηφίσετε αυτές τις συμβαστικές λύσεις τα υπόλοιπα θα ξεπεταχθούν πολύ γρήγορα. Ο καθένας φυσικά ψηφίζει όπως θέλει, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλές συμβαστικές λύσεις και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για τις καρποφόρες διαπραγματεύσεις μας. Ευχαριστώ αλλά η ποιότητα πιο σημαντική από το χρόνο. Ο Ιβο Μπέλδοτ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτό το τελευταίο που είπατε. Ας ε, συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Πολύ καρποφόρα, πολύ υποδομητική η προσέγγιση του και οι προτάσεις του. Υποστηρίζουμε όλες τις συμβαστικές που μας προτείνατε τις περασμένες εβδομάδες. Αναφερθήκατε στους βασικούς ε, βλεκόμενους φορείς ICO e και IMO είναι ε, φιλόδοξες οι κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες έχουν καταλήξει αυτά τα θεσμικά όργανα, κυρίως αυτό που λέμε πως ε, ζητάμε και απαιτούμε ρητά μέχρι το πέρας του 2016 να καταλήξουν σε ένα αξιόπιστο εργαλείο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μειώσεις στις εκπομπές. Η τροπολογία 4, η συμβαστική 4, είναι η πεμπτουσία αυτής της έκθεσης και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, διότι μιλάμε για την αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και για τους ε, διάβλους ε, κατανομής ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή για τις οδικές μεταφορές και για την αποθήκευση αυτού στη συμβαστική 6 μιλάμε για την προώθηση των εναλλακτικών πηγών, βιοαέριο και το καθεξής. Τέλος πάντων, για να μην τα λόγο, θα ήθελα να κάνω ίσως δύο επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Χρειαζόμαστε άλλο ένα στόχο πρόσθετο για το 2030 για τις μεταφορές. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Έχουμε ένα γενικό στόχο, μπορεί κάποιος να, να συζητά για τη δυνατότητα να έχουμε υποστόχους. Ας έπεται όμως και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, κατανομή των βαρών ε, για τον ETS, οπότε για την, ε, τα δικαιώματα εκπομπών ρήπων δηλαδή, οπότε θα έπρεπε ίσως να περιμένουμε. Ε, σε σχέση με μια τροπολογία ε, υπαριθμών 36 των σοσιαλιστών ε, θα έπρεπε να την υποστηρίξουμε, μιλάμε για τον Κοπέρνικο, για τις, τα προγράμματα γεωπαρατήρησης. Αυτά συμβάλλουν στα προγράμματα καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και μας ικανοποιεί η συμβατική πρόταση στην οποία καταλήξαμε και προτείνω να την ε, υπερψηφίσει η Επιτροπή και ευχαριστώ και τους σκιώδες. Ε, ευχαριστούμε η Κριστίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδες σε πολύ επικοδομητική δουλειά που κάναμε. Και νομίζω ότι αυτή η συλλογική δουλειά θα πρέπει να συνεργαστεί. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία εξέδωσε γνωμοδότηση η Επιτροπή μα είναι σημείο αναφορά σε σχέση με τι προτεραιότητε Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη και τη συνόδου του, στο Παρίσι τη COP21. Νομίζω ότι υπάρχει συμβασμό σε σχέση με το να στείλουμε ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα ότι ε, χρειαζόμαστε δεσμευτικού στόχου και ε, επιδιώκουμε ε, ο τομέα των μεταφορών να είναι στον πυρήνα των προσπαθειών για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό όχι μόνο μόνο ε, στο πρωτόκολλο του Παρισιού, το κεντρικό έγγραφο, αλλά και στο θεματολόγιο των λύσεων τη COP21 για να προταθούν συγκεκριμένε πρωτοβουλίε και να ε, τονίσουμε ε, ποια είναι η ευθύνη και των μη κυβερνητικών εμπλεκομένων φορέων πέρα από την κινητικότητα, γιατί ξέρουμε ότι το 1 τέταρτο των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών είναι σε μια αστικές περιοχέ. Στη συνέχεια το Ταμείο για το Κλίμα, να άλλη μια ιδέα που θελήσαμε να προωθήσουμε για να συμπληρώσουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όμως υποτιμά τη σημασία αυτή τη βασική πρόκληση τέλο. Ε, Υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να καταθέσει φιλόδοξες ε, νομοθετικές ε, προτάσεις ούτως ώστε το, κλίμα, το πακέτο κλίμα ενέργεια για το 2030 να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν και να σημειωθεί και πρόοδος για τις εκπομπές των αυτοκινήτων. Σας ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συμβαστική λύση και θα τις υποστηρίξουμε αύριο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή, τους εισηγητές για το έργο τους για αυτό το θέμα. Αλλά οι τροπολογίες συμβασμού οι οποίες έχουν κατατεθεί δεν υποστηρίζονται από την ομάδα μας. Η ομάδα μας θα καταψηφίσει αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος η Μάισνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ φυσικά θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Κάνανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας και έχουν βρει πολλές ε, συμβαστικές τροπολογίες που μπορούν να υποστηριχθούν από την ομάδα μας, από την Άλντε και έχουμε ελάχιστες τροπολογίες που έχουμε καταθέσει πέραν των συμβιβαστικών Επομένως, εμείς χαιρόμαστε για το γεγονό ότι έγιναν δεκτές οι δικές μας για τη συμβαστική ένα είναι φανερό ότι πρέπει να γίνει πιο ορατός ο τομέα των μεταφορών και να εργαστεί για μια βιωσιμότερη μορφή μεταφορών σε σχέση με, τις, ε, με το περιβάλλον και όπως είπατε προηγουμένως η ΚΑΟ και η ΙΜΟ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους σε Διεθνέ επίπεδο για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί στο προσκήνιο. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Στην τροπολογία 3 αφορά πάλι στη μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών και να έχουμε μια επιμελητία μεταφορών που να είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη συνέχεια έχουμε τη συμβασική τροπολογία για τα εναλλακτικά καύσιμα τροπολογία συμβασμού 5 αφορά την κοινή ναι. κινητικότητα που λαμβάνει υπόψη και τις δημόσιες μεταφορές. Για την έκτη αφορά το μείγμα ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και η τροπολογία αυτά στην σωστή, στο θεμητό ανταγωνισμό και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που φυσικά παίζουν σημαντικό ρόλο για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία φιλική με το κλίμα. Είμαστε λοιπόν πολύ ικανοποιημένοι από τις διαπραγματεύσεις και προσβλέπουμε στους νέους δεσμευτικούς ε, στόχους. Υπήρξε διαφορά εδώ μεταξύ των ε, ε, πολιτικών ομάδων και εκεί πέρα πρέπει να ψηφίσουμε χωριστές τροπολογίες και εγώ θέλω να παραπέμψω σε μια συγκεκριμένη τροπολογία όπου αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν διεθνώς δεσμευτικοί στόχοι. Εάν δεν γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την δική μας ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό <clears throat> επίπεδο. Αυτό για την τροπολογία 40. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τους συζητητές για την καλή συνεργασία. Η Μαΐα Κίλανεν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστώ τον κύριο Έκχαρτ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Εμείς πρώτη να συμφωνήσουμε όλους τους θεσμούς που Και επίσης θα πρέπει να δούμε όμως και κάποια άλλα ζητήματα. Μια από στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο προέχει είναι να μπορέσουμε να καθορίσουμε το τι πρέπει να γίνει για το περιβάλλον. Θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι ή ουραγοί. Τι κάνουμε τη σημερινή μέρα. Προσέχουμε κάποιες τεχνολογίες που μπορεί να διευκολύνουν, αλλά από την άλλη μεριά φερόμαστε κάπως εγωιστικά, διότι δεν απαιτούμε να αλλάξει η συμπεριφορά των Χριστών, του κόσμου. Τα πράγματα αλλάζουν. Οπότε θα πρέπει να δούμε κάποια εναλλακτική τεχνολογία. Ας πούμε την ασύρμενη τεχνολογία. Διάβασα το συμβαστικό κείμενο του κυρίου Έκχαου και αυτό μου θύμισε κάτι που είχε πει ο Χένρι Φόρντ Και λέει ότι αν ρώτηκε τον κόσμο τι επιθυμεί, τότε θα του απαντούσαν πιο γρήγορα άλογα. Βέβαια ο κόσμος τώρα ίσως έβαλε μυαλό. Και ίσως ε, η επιθυμία είναι τώρα για φρέσκα, καινούργια άλογα. Και όχι απλώς πιο γρήγορα αυτοκίνητα. θα το σκεφτούμε. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην Κομισιόν ο Μάρτιν Βέστροπ για την ε, DG Energy. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως, α. Όπως είπατε, η Ενεργειακή Ένωση είναι μια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μας απασχολήσει ως προτεραιότητα την επόμενη διετία και ελπίζουμε ότι θα τύχουμε τις πλήρους υποστήριξης για αυτήν την στρατηγική, γιατί αμέσως να τις ε, διακοπέ σε μια ψηφοφορία αλλά και στην Ολομέλεια. Οπότε θα μπορέσουμε και εμεί να προχωρήσουμε στην εφαρμογή τη στρατηγική. Όπω ξέρετε, έχουμε πρωτοβουλία στην από την εβδομάδα για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με το ότι το σχέδιο κειμένο της ίτρε δεν έχει θίξει τα θέματα μεταφοράς. Γι' αυτό ακριβώς και σας ευχαριστούμε πολύ που αποφασίσατε να προχωρήσετε σε μια δική σας ονομαδότηση. Είχαμε συμφωνήσει όταν την παρουσιάσατε, θεωρούμε ότι βελτιώνουν τα πράγματα οι τροπολογίες και περιμένουμε αναγνώριση την αυριανή ψηφοφορία. Και βέβαια θα γίνει και στην Ήτρα η αντίστοιχη ψηφοφορία. Τώρα κάποια επιμέρου σημεία, βεβαίω και συμφωνούμε 100% ε, ότι οι μεταφορές είναι τομέας πάρα πολύ σημαντικός. Στον αφορά την εξάρτησή μας από τις και εξαρτήση κανονικά όσον αφορά τα τα καύσιμα πρόκειται να αυξηθεί στο μέλλον. Βέβαια, τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν σε περισσότερες εκπομπές διοξιδίου, όπως είπατε, και άρα χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, ούτως ώστε να συνεχίσουμε την μείωση στο μέλλον αυτών των εκπομπών. Είναι σημαντικό, όπως είπατε, το να δούμε τους διαφορούς τρόπους μεταφορών στην Ένωση. Να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους τρόπους μεταφορών που είναι πιο αποτελεσματικά. Να αναβαθμίσουμε τις ανεωσμένες πηγές ενέργειας. και τον εξυλογητισμό των διαφόρων τρόπων μεταφορών και, τις, και να δούμε τι θα γίνει με, την, με τον εξελικτισμό της κινητικότητας όπως αναφέρθηκε. Οπότε ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον προς την πρωτοβουλία μας και βλέπουμε στην αυριανή ψηφοφορία πρόεδρος. Ο κ. Μέτκα από την ε, Move. Ε, εδώ είμαι, ναι, ναι. Κα... Και εμείς Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο και βλέπω ότι ευθυγραμμίζεστε σε μεγάλο βαθμό με τις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μοναδικό σχόλιο που θέλω να κάνω είναι πως στην COP21 και τη Διεθνή Διαπραγματεύση που θα γίνουν για τις μεταφορές αυτό που θα έχει σημασία είναι προς τον ε, ΙΚΑΟ και τον ΑΕΜΟ να στείλετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα με ε, καταληκτικέ ημερομηνίε. Πότε πρέπει δηλαδή να έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους εργασίες. Εμείς από πλευράς μας ήμασταν ξεκάθαροι για αυτό το θέμα στην ανακοίνωσή μα. Πέραν αυτού, Είμαστε ικανοποιημένοι και με ηλεκτρικά μέσα θα πάμε στην COP21, ε, εκτός από αυτούς που θα πάνε με ποδήλατο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τελευταία σας φράση. Και τώρα θα δώσω και πάλι το λόγο στους δύο εισηγητές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλύψαμε τα περισσότερα από τα σημαντικά ζητήματα και η σημαντικότερη πρόκληση είναι ότι το 94% ε, κατά το 94% εξαρτώμαστε από το πετρέλαιο παρότι υπάρχουν ε, άλλες διαθέσιμες πηγές ενέργειας και άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο μετάβασης ε, σε πιο βιώσιμες αστικές μεταφορές. 70% των Ευρωπαίων ζουν σε αστικές ζώνες. Άρα ε, το χωροταξικό μας σχεδιασμό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να αναλαμβάνονται ένα και περισσότερο πρωτοβουλίες όπως ποδηλατόδρομοι και το καθεξής για να ε, καταστεί περισσότερο βιώσιμη η μετακίνηση να μειώσουμε στις εκπομπές Λοιπόν, Πολλοί μίλησαν για τα ηλεκτρικά οχήματα. Πέρα από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα όμως έχουμε και το θέμα πώς θα πρέπει να είμαστε ενεργειακά ουδέτεροι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές εναλλακτικέ λύσεις, ε, καύσιμο που βασίζονται σε υδρογόνο, ηλεκτροκίνητα, οχήματα. Για τον περιορισμό των εκπομπών δεν έχουμε μία μόνο λύση και στις θαλάσσιες και τις νερές μεταφορές επίσης έχουμε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις και θα πρέπει αυτό να συνυπολογιστεί σε διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό για την Ευρώπη να καταλήξει σε συμφωνία και για τα δύο. Δεν θα πρέπει η Ευρώπη μόνη της να υπομειστεί την ευθύνη για την βιώσουμε αυτή τη συνέργεια. Και μην ξεχνάμε ότι τίθεται και μείζον ζήτημα ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε πάντω ε, για τη συνεργασία και Ελπίζω αύριο να υποστηρίξει η Επιτροπή συμβαστικές προτάσεις. Σας ευχαριστούμε και τώρα ο Μπασίκου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους σκιώδους εισηγητές για τη συμβολή τους. Νομίζω ότι δεν θα, δεν είναι άνευ περιπλοκών η αυριανή ψηφοφορία και βλέπω ότι δηλώνει ικανοποιημένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θέλω μόνο να τονίσω πως ξεκάθαρα εμείς ζητάμε από την Επιτροπή μέσα στην έκθεση, όχι γενικότερα για το COP21, αλλά για το τομέα των μεταφορών να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε ε, αποτελεσματικότητα, αλλαγή μοντέλο, η ε, αποφυγή κάποιων μεταφορών, καθώς και περιορισμός τελάχιστο των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι μέρος της COP21 και ζητάμε μετά από το Παρίσι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή το επόμενο βήμα και να καταθέσει ένα πακέτο συγκεκριμένα για τις μεταφορές. Το έχει αποδείξει το μέσο ότι αξίζει ε, ιδιαίτερη νομοθετική προσοχή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και νομίζω ότι εφόσον είσαστε τόσο ικανοποιημένοι, καλά θα κάνατε να ακολουθήσετε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο για το δρόμο μέχρι το Παρίσι, αλλά και μετά. Αύριο θα ψηφίσουμε, αύριο πρωί, γνωρίς. και στην Ήτρε 22 και 23 Σεπτεμβρίου, στην ΕΜΒΗ 22 Σεπτεμβρίου και μετά Ολομέλεια. Επόμενο σημείο, προπολογισμό 2016, ο Μαρτιμιλιάνο Σαλίνη είναι ο εισηγητή μα. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα, ας ε, θυμηθούμε ποια είναι τα σοβαρά, τα, τα, τα πιο σημαντικά ορόσημα που έχουν μπροστά μας, γιατί έχουμε ε, τις ε, τροπολογίες για τι οποίε ισχύει η, η τη της 22ης ε, Ιουλίου και όπω ξέρετε οι συνάδελφοι οι τροπολογιστέ αφορούν την γνωμοδότηση που θα κατεβάσουμε ή το σύνολο του προπολογισμού. Υπάρχει μόνος ε, η δυνατότητα αλλαγών. Και μεταξύ αυτών των προπολογιών έχουμε επίσης και κάποια πιλωτικά προγράμματα. Είναι αυτά ε, τα οποία έχω ξεχωρίσει 12. Οπότε ακριβώς αυτό θέλουμε να πετύχουμε με αυτή την ε, διαδικασία και έχουμε την προθεσμία της 22ης Ιουλίου. Τώρα, 31 Αυγούστου είναι η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση. Κατόπιν θα διαβάσουμε και ονόμα στον κύριο Φερνάντες. που όπως ξέρουμε από εκείνη την ακρόαση είναι ο γενικός εισηγητής. Τώρα, στις λεπτομέρειές τους, μπορούμε να πούμε ότι ο πυρήνας της γνωμοδότησης αναφέρεται στα καινοτόμα στοιχεία τα σχετικά με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, δηλαδή στο πλάνο Γιούγκερ. Οπότε αυτό είναι στην καρδιά του προπολογισμού μας. Η δε πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ε, αρκετά ετολμηλή, γιατί είχαμε πει ότι έχουμε τα 8 εκατομμύρια τα οποία είχαμε ζητήσει και ήθελαν να καλυφθεί το Horizon και το Connecting Euro Facility. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις σκληρές και αλλάξαμε την, ε, την πρικοδότηση και είπαμε, πήγαμε στα 5 εκατομμύρια συν 1 για το ΣΕΦ. και είπαμε ότι έχουμε τα 55 εκατομμύρια ε, για το ΣΕΦ, ε, το Connecting Europe, το οποίο θα αφορούσε μόνο τις μεταφορές και όχι και τηλεπικοινωνίες. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί η πανίδαση εκεί θα μπορούσε να επιφέρει αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τις επενδύσεις από πλευράς κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Και πέραν επομένως, του οικονομικού θέματος έχουμε το θέμα των επιδοτήσεων. Και είπαμε ότι έχουμε τις με μεταφορές, εσωτερικές πλωτές και οπότε εκεί βλέπουμε ότι ο ρυθμός των επενδύσεων είναι εδώ βραδύτερος από ό,τι άλλο. Άρα γι' αυτό και είπαμε ότι κάτι να γίνει τώρα με το ΕΦΣΙ. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί στη θέση μας. Αλλά πέραν αυτού υπάρχει το άλλο κεφάλαιο που αφορά τη σχέση του προπολογισμού με το σύμφωνο σταθερότητας. Γιατί τα 28 κράτη-μέλη έχουν πει ότι σε αυτή τη φάση δεν βοηθά το σύμφωνο σταθερότητας για κάποιες ε, επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην τόνωση της οικονομίας της Ευρώπης. Από τη βγαίνουν οι επενδύσεις από το δημόσιο χρέος, τον υπολογισμό του. Όμως έχουμε τελικά κάποια πιο στενή ερμηνεία των σχετικών αριτρών. Και είπαμε ότι θέλουμε εδώ να καλύψουμε τους βασικούς πυλώνες της Επιτροπής μας της ε, πολιτικής μας όπως τα, τα, τα TNT, τα ευρωπαϊκά δίκτυα για τις μεταφορές. Να καλύψουμε λιμένες, αερολιμένες, όλα αυτά είπαμε ότι είναι τα κλειδιά για περισσότερη ανταγωνιστικότητα, άνοιγμα προς τον κόσμο και έχουμε το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Και σχετικά με αυτό έχουμε πρώτα τη σχέση μεταξύ των εθνικών αρχών για την ασφάλεια και των Σιδηροδρομικών αρχών της Ευρώπης. Και σε δεύτερη φάση είναι το RTMS σαν ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ε, πολιτική αεροπορία, το focus που θα παρέχει εγγύησεις για ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και προστασία των ε, δικαιωμάτων των ε, πολιτών. Αλλά είναι και το θέμα του τουρισμού, σε σχέση και με αυτά τα έργα, τα projects που έχουν προταθεί και είπαμε ότι για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να καλυφθούν αυτά τα projects και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας οριζόντιος γραφείος, οριζόντια αρμοδιότητα πολλών επιτροπών. Τέλος δε, καλύψαμε εδώ αυτήν την μνήμα που θέλαμε, αυτό το οποίο ήθελε η συνάδελφος Κούνεν όσον αφορά αστικές μεταφορές, γιατί πάνω από το μισό πληθυσμό παγκοσμίω και πάνω από 70% των Ευρωπαίων ζουν στις πόλεις. Αλλά θέλουμε να έχουμε αστικές ε, επικοινωνίες οι οποίες να είναι αποτελεσματικές και αυτό θα βοηθήσει γενικότερα παντού την ανάπτυξη πρόεδρος. Πυρίτσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σελήνη για την πολύ καλή θέση του για το σχέδιο προπολογισμού του 2016. Έχουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίσης και τη θέση του Συμβουλίου. Έτσι μπορούμε να προτείνουμε βελτιώσεις και να ζητήσουμε και ε, πρόσφορες γραμμέ ε, στον προπολογισμό που θα ταιριάσουν με τις προτεραιότητε στον τομέα των μεταφορών. Η πρώτη διορθωτική επιστολή για το σχέδιο 2016 αυξάνει ε, τις επιστώσεις άλλες υποχρεώσεων ε, για το ΣΕΦ βάσει και των δεσμεύσεων του ΕΦΣΥ ε, καθώς και αυξάνει και τις πρώτες δεσμεύσεις που αναλάβει στα πλαίσια πάλι του ΕΦΣΥ για το ΣΕΦ. Όμως το Συμβούλιο προτείνει περικοπές ε, στις επιστώσεις και πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων και δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ενημερωθήκαμε για την, το ανεπροηγουμένο ενδιαφέρον που υπάρχει υπάρχει στον τομέα των μεταφορών στο ΣΕΦ. 681 επιλέξιμες προτάσεις έχουν κατατεθεί, μόνο οι 276 τελικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το ΣΕΦ και άρα χρειαζόμαστε και κατάλληλη χρηματοδότηση. Άρα οι προβλεπόμενες πιστώσεις, ε, ανάλυση υποχρεώσεων και πληρωμών ε, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να τηρηθούν. Επίσης, ε, στο, το Συμβούλιο προτείνει περικοπέ για το ε, ε, προηγούμενο πρόγραμμα των διασυνοριακών δικτύων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την περικοπή του Συμβουλίου, διότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεξόφλητων λογαριασμών. Δεν διοχετεύει του απαιτούμενου πόρου του Συμβούλου για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του οργανισμού. Προτείνονται περικοπέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολλού και σημαντικού οργανισμού. Δεν μπορούμε. Ε, να συμφωνήσουμε με τις περικοπές ενός εκατομμυρίου και άνω ε, σε οργανισμούς που είναι βασικά αρμόδιοι για το ΣΕΦ και για το συντονισμό των προγραμμάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην απαλλαγή για το 2013 έχει τονιστεί ήδη του οργανισμό χρειάζεται ο πετούμενο ποσό, ώστε ικανοποιητικά να μπορέσει να ανταποκριθεί στι δεσμεύσει που έχει αναλάβει και τα καθήκοντα που το έχουν ανατεθεί χρειάζονται οικονομική και ανθρώπινη πορεία. Επίση, θέλουμε να αποκατασταθεί η αρχή πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το σιδηροδρομικό ε, οργανισμό, διότι θα αυξηθούν ε, μετά την έγκριση του τετάρτου σιδηροδρομικού πακέτου οι αρμοδιότητε αυτού του οργανισμού και δεν θα είναι σε θέση ο οργανισμό λοιπόν να ανταποκριθεί μόνο με του φόρου που προέρχονται από του από του φόρου και από τα τέλη. Επίση, χρειαζόμαστε μια νέα γραμμή για τον τουρισμού αυτό έχει καταχειρηθεί. Όμω, για τα προγράμματα που σχετίζονται με τον τουρισμό θα χρειαστεί χρηματοδότηση από διαφορετικέ γραμμέ του προϋπολογισμού και γι' αυτό χρειάζεται συντονισμός ε, για να διοχετεύονται πορεία από δύο διαφορετικέ πηγέ. Επίση, για τι δράσει και τα πολιτικά προγράμματα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προγράμματα σε αυτό το τομέα. Τέλος, αλλά σημαντικό είναι ο ρόλος ε, της έρευνας, ε, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη σημασία της έρευνας στον τομέα των μεταφορών, κυρίως ε, ακολουθώντας τον, ε, έναν δρόμο προς ε, ευφιέστερα συστήματα μεταφορών για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές. δεν μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε με τις προτινόμενες από το Συμβούλιο Περικοπές στον τομέα της έρευνας για τις μεταφορές κατά πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα εγώ θα καταθέσω τροπολογίε ώστε να αποκατασταθούν οι πιστώσεις που υποχρεώσεων και πληρωμών και να αντιταχθούμε στις περικοπές που προτείνει το Συμβουλίο. Ευχαριστώ τον Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Έχω πολλά σχόλια. Πρώτα απ' όλα το σχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν. Γενικά δείχνει μια μικρή αύξηση πάνω από τον πληθωρισμό. Μπορεί να θεωρήσει κανείς λοιπόν ότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι λογικός σε ό,τι αφορά το ύψος του. Όμως, όμως όπως ελέγχθη, υπάρχουν ορισμένε πτυχέ που πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Ο λειτουργικό φορέα καταρχήν για τα δίκτυα βλέπει να μειώνεται η χρηματοδότησή του τη στιγμή που θα έπρεπε να λειτουργήσουν όχι μόνο αυτά τα 13,4 δισεκατομμύρια από τα επιλεγμένα σχέδια, αλλά πρέπει να κάνει και μια νέα πρόσκληση ενδιαφέροντα στο τέλο του χρόνου. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να μειωθούν τα λειτουργικά κονδύλια αυτού του φορέα, ο οποίο ήδη δεν είχε πάρα πολλά χρήματα στη διάθεσή του. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό τη Κομισιόν, η μείωση του προπολογισμού έρευνα είναι ουσιαστικά απαράδεκτη όταν υπάρχει μια διάβρωση του προϋπολογισμού, αλλά αυτό θα οδηγήσει και σε μια καθυστέρηση της εφαρμογής των προγραμμάτων που θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγάλες <clears throat> ανησυχίες σε εμάς, ιδίως για, τα, για τις κοινέ συμπράξεις, τα joint undertaking. Επίσης η μείωση της χρηματοδότησης του Γαλιλαίου και σε πιστώσεις πληρωμών και υποχρεώσεων για 5,66 αυτό για ένα σχέδιο το οποίο είναι σε φάση ανάπτυξης και ήδη αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, αυτό θα είναι πολύ αρνητικό. Και τέλος, για τους αποκεντρωμένους φορείς, η Κομισιόν επιμένει στα, στο πλαίσιο του πολιετούς προϋπολογισμού. Εμείς δεν θέλουμε να μειωθούν οι πόρτες σε ασά του ε, φορέα θαρασιών θεμάτων και του τομέα για τα συνδρομικά, ε, θεωρούμε ότι η Κομισιόν επιμένει και πάλι να μειωθούν τα οργανογράμματα σε αυτούς τους ε, ε, φορείς παρά το γεγονός ότι μόνο το 1 τέταρτο του προπολογισμού τους καλύπτει. Λοιπόν, η Κομισιόν έρχεται σε αντίφαση με τις πολιτικές κατευθύνσεις και συγχρόνως περιορίζει το προσωπικό φορέων που έχουν ήδη δικό τους, ε, δικού τους πόρους και επομένως πρέπει να χαράξουν μια αυτόνομη πολιτική προσωπικού. Αυτό για μένα είναι ακατανόητο. Και τώρα σε ό,τι αφορά τη θέση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο γενικά αφαιρεί, μειώνει τα κονδύλια που θέτει η Κομισιόν και φυσικά μετά οδηγείται σε μια απόφαση κατά ομοφωνία. Πολύ σπάνια όμως βλέπει κανείς το Συμβούλιο να αυξάνει ακόμα περισσότερο τις περικοπές που προτείνει η Κομισιόν και αυτό θα μας φέρει σε ένα σημείο όπου ουσιαστικά δεν θα μπορούμε να συμπληρώσουμε τον τέταρτο πυλώνα, τον τεχνικό πυλώνα. Για το σχέδιο τώρα προϋπολογισμού σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμίζεται με αυτά που διαπραγματευτήκαμε το Δεκέμβριο με το Συμβούλιο. Να θυμηθούμε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο θα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα του χρόνου για την ενδιάμεση μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου για τα περιθώρια. Γιατί τα 2,4 δισεκατομμύρια τα οποία διεσώθηκαν από τα νύχια του Συμβουλίου για το Connecting Europe Facility είναι το μέγιστο που μπορούμε να δεχτούμε ως ποσό αφαιρούμενο από αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει. Κάθε χρόνο λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε με ένα αγώνα για να μην χάσουμε περισσότερα από εσά στον τομέα αυτό. Αν αναλύσει κανείς λοιπόν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, εκεί έχουμε πετύχει να να πάρουμε κάποια χρήματα από το περιθώριο του τρέχοντος έτους. Αυτό λοιπόν έχει γίνει και το 2014 και το 2015. Αυτό δείχνει ότι αν έχουμε μια στεναρή θέση και του χρόνου μπορούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις περικοπές του Συμβουλίου. Και κλείνω λέγοντας ότι κάθε χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά τις πιστώσεις μεν, αλλά αφορά και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά σχέδια. Έχουμε πολλά πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις κάθε χρόνο, περισσότερα φυσικά από τη χώρα στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να γίνουν επιλογές μέσα στα πλαίσια αυτά. Εγώ θα προτιμούσα η Επιτροπή μας να κάνει κάποιες επιλογές να μην φτάσουμε σε μια θέση που θα αναγκάσει την Κομισιόν να κάνει αυτή τις επιλογές αντί για μας. Και σας παραπέμπω και στην έκθεση της Τεχνικής Επιτροφής της Κομισιόν που σε επόμενες 48 ώρες θα θέσει σε μια ιεράρχηση τα σχέδια αυτά. Και νομίζω ότι η σωστή μας στάση εδώ θα ήταν να υπερασπιστούμε τις θέσεις του προπολογισμού που έχουμε υποστήριξει στο παρελθόν και ακολουθώντας τη βασική μας αρχή να βοηθήσουμε την Κομισιόν και να αντισταθούμε στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Η Μάια Κίλωνεν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σαλίνη για τα τόσα ωραία που μας εξήγησε. Εγώ όμως θέλω να τονίσω πόσο σημαντική υπόθεση είναι το θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Θα πρέπει εκεί να εκφράζουμε την άποψή μας πιο δυναμικά, όχι με μια απλή σύσταση. Η το πλευρά ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας είναι υπόθεση σημαντική στην Ευρώπη. Ε, απασχολούμεθα με αυτήν την υπόθεση χρόνια, χωρίς να καταλήξουμε κάπου. Και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε τους ε, στόχους μας για τους ε, Ευρωπαίους και μη επιβάτες. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεμερίσουμε το θέμα τόσο γρήγορα, τόσο συνοπτικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα κονδύλιο σχετικό με τον τουρισμό. Και αυτό μας έχει υποσχολήσει πολύ καιρό στην Επιτροπή μα, αλλά τελικά δεν έχουν διατεθεί αρκετά κονδύλια για τον τουρισμό. Επομένως, ε, θα ήταν σωστό αυτό να καλυφθεί. έτσι ο τουρισμός να μπορέσει να βοηθήσει γενικότερα. Κάτι άλλο το οποίο αφορά την λευκή βίβλο για τις μεταφορές. Έφτασε αργά, οπότε δεν υπήρξε ο χρόνος να μπορούσαμε να το μελετήσουμε και να καταλάβουμε κάποιες τροπολογίες. Τι γίνεται με την ε, πολιτική μας για την Αρκτική, και τις μεταφορές. Τι γίνεται με το ότι διαφέρει πάρα πολύ σκανδιναβικές χώρες. Μήπως θα ήταν δυνατόν και αυτό το θέμα να μπει στις προτεραιότητες. Δεν το προσέξαμε όσο χρειαζόταν. Ευχαριστώ. Δεν είναι πρόβλημα βέβαια στην αρκτικό κύκλο η κλιματική αλλαγή γιατί κάνει πιο εύκολες μεταφορές και όχι πιο δύσκολες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Σαλήνη Πρόεδρε για το έργο του. Θα κατεβάσουμε κάποιες τροπολογίες προς αυτές τις ε, κατευθύνσεις κυρίως όσον αφορά το θα πρέπει να έχουμε περισσότερη διαφάνεια Τα είπαμε και με την ε, Επίτροπο την περσμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει για όλα αυτά τα έργα, τα σχέδια να υπάρξει διαφάνεια. Για όλα αυτά τα οποία πρότεινε, για αυτά για τα οποία έχουμε κάποια εκταμείευση πόρων. Την μεγίστη δυνατή διαφάνεια. Αυτά θα προτείνουμε. Για τη χρηματοδότηση, για του χρηματοοικονομικού μα πόρου. Όλα αυτά θα πρέπει να περιβάλλονται από νομιμότητα. Και έτσι να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από όλα αυτά τα κουσούρια τα οποία μαστίζουν τη χρηματοδότησή μας. Τώρα όσον αφορά την περιβαλλοντική επίπτωση των ε, έργων και σχεδίων, αυτό θα πρέπει να γίνει τόσο γίνεται καλύτερα, πιο καλά δηλαδή. Αυτά λέτε δηλαδή που χρηματοδοτούμε, πώς επιδρούν στο περιβάλλον. Τελευταίο, αλλά σημαντικό, να δούμε κάτι σε σχέση με τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα πρέπει πάντοτε να τους έχουμε υπόψη. Όποτε θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα μεγάλο έργο υποδομής. Και να μην ξεχνούμε ότι ακριβώ οι υποδομές είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Να μην ξεχνούμε αυτό το οποίο επιθυμούν οι Ευρωπαίοι για αυτά τα έργα που εμείς θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Πριν να αφουγκραστούμε τον πολίτη. Κριστίνη σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή για την παρουσίαση που μας έκανε σήμερα. Δεν έχει από πολλούς συναδέλφους μου, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι, ότι μεγάλη ικανοποίηση βλέποντας ότι στο σημείο 2 αναγνωρίζεται ο ειδικό χαρακτήρα ορισμένων φορών μεταφορών, ιδιαίτερα των συνδρομικών μεταφορών που πρέπει να έχει περισσότερε επιδοτήσει και όχι μονάχα χρηματοδοτικά εργαλεία και επίση αναφέρθηκαν στην αδελφή μου στον προπολογισμό της ΕΡΑ, του Σιδηροδρομικού Φορέα. Μόλις τελειώσαμε τον τρίλογο για την τεχνική πτυχή και βλέπουμε ότι το προσωπικό ε, μειώνεται κατά δύο υπαλλήλους ενώ χρειάζεται να ενισχύσουμε τους πόρους αυτού του φορέα και είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε το να διατηρήσουμε τον προπολογισμό αυτού του φορέα <clears throat> και να διατηρήσουμε το προσωπικό αυτό. Πηγαίνει επέκεινα της Επιτροπής Μεταφορών. Θα πρέπει να πείσουμε όλους τους συναδέλφους μας της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής που δεν μας ακολουθούν πάντα για τα θέματα αυτά. Και η δεύτερη παρατήρησή μου για το πρόγραμμα ε, της ε, Ευρώπης 2020. Αναφέρθηκε αυτό, του ορίζοντα 2020 μάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα και στον ε, επερχόμενο προεπολογισμό ο οποίος θα παρουσιαστεί και θα φυσικά καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ισαμπέλα Ντεμόντε. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, γνωμοδότηση που είναι τόσο πλήρης για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν ε, τις μεταφορές. Αλλά επίσης έχει καλύψει και το θέμα του τουρισμού. Το αν δούμε τι γίνεται με το Connecting Euro Facility. Εκεί είχαμε το αρνητικό φαινόμενο των περικοπών. Γιατί ακριβώ τώρα έχουμε το Ταμείο Γιούγκερ και άρα δεν θα πρέπει να μειωθούν οι ε, υποστήριξη, οι δυνατότητες που υπάρχουν για το ΣΕΦ να δούμε τι μπορεί να γίνει για τις ε, υποδομέ και έχει δίκιο ο εισηγητή ότι δηλαδή ίσως χρειάζεται τώρα να γίνει επίκληση κάποιων επιδοτήσεων. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με την κινητικότητα στις πόλεις. Ε, το συζητήσαμε εδώ και είπαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει ο σχετικό προγραμματισμό για τις ε, μεταφορές στις πόλεις. Να δούμε πώς θα γίνουν πιο αποτελεσματικές αυτές οι μεταφορές. με τον προγραμματισμό θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην χρήση των οδών και όσον αφορά την χωροταξία στις πόλεις και τελικά θα καταλήξουμε να έχουμε ε, λιγότερα μποτιλιαρίσματα. Άρα προγραμματισμός και χωροταξία για τα μέσα επόμενα χωριά, τα επόμενα χρόνια, οπότε θα διορθώσουμε το πρόβλημα που ήδη υπάρχουν τώρα θα ήθελα να σας πω ότι όπως είπαν οι συνάδελφοι χρειάζεται ο τουρισμός ένα κονδύλιο γιατί είπαμε ότι έχουμε κάποιους πόρους διευθύνται άμεσα άλλους έμεσα αλλά δεν επαρκούν θα πρέπει να είναι η προσβασιμότητα εύκολη σε αυτούς τους πόρους και μην υπάρχει μια κατάτμιση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης. αλλά χρειάζεται και η Επιτροπή να κάνει μια ανακοίνωση σχετικά. Μια που ο κλάδος του τουρισμού επιδρά πάρα πολύ ε, εκεί όπου υπάρχει αυτή η δραστηριότητα, που αναπτύσσεται αυτή η δραστηριότητα και θα πρέπει να μην έχουμε κοινωνικό dumping. Χρειάζεται επομένω λοιπόν να προσέχουμε τον τριτογενή τομέα και αυτό να γίνει με συγκεκριμένα κονδύλια. Η κρίση έχει χτυπήσει και τον τουρισμό. Να δούμε τι θα γίνει επομένω τα μέσα σε επόμενα χρόνια. Θα το συζητήσουμε αυτό και αύριο. Αλλά ο βασικός ε, ιστός εδώ, ο είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει τη χώρα μα Πρόεδρος. Η κυρία Μάισνερ, πάρα πολύ σύντομα. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πολύ σωστά ο εισηγητής υπεγράμμισε το γεγονός ότι το Connecting Euro Facilities έχει χάσει πάρα πολλά χρήματα τα οποία πήγαν στο EFCI, EFSI μάλλον. Ένα μεγάλο μέρος των ε, επενδύσεων μπορεί να έρθει στον τομέα μεταφορών, αλλά θα πρέπει εμείς να κάνουμε τα απαραίτητα ως Επιτροπή Μεταφορών να εξασφαλίσουμε ότι όσο δυνατόν περισσότερα από τα χρήματα θα παραμείνουν στο Connecting Eurofacility Facility και θα βρεθούν άλλες λύσεις για να χρηματοδοτηθεί το EFSI. Αυτό ήθελα να το ε, αναφέρω και αφού είναι και ο πρώην πρόεδρος μας εδώ ήθελα να το πω οπωσδήποτε. Για την Κομισιόν. Η κυρία Αμπαγαρότε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που με έχετε καλέσει εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών Κομισιών. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον κύριο Σαλίνη για το σχέδιο γνωμοδότησης και καταγράφει τα σχόλια τα οποία διατυπώθηκαν. Η Κομισιόν θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στην πολιτική μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΦΣΙ έχει πάρει χρήματα βέβαια από το Connecting Europe Facilities αλλά πιστεύουμε ότι πολλά σχέδια μεταφορών θα συμπεριληθούν στο ΕΦΣΥ και επομένως αυτό θα οδηγήσει σε αντίστοιχη χρηματοδότηση για τις μεταφορές. Αναφερθήκατε στο ERTMS, στους ενιαίους ουρανούς, τις διατροπικές ε, συνδέσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία τα λαμβάνουμε υπόψη μας και εγώ συμμερίζομαι την απόψη του κύριου Πυρίνσκη και του κ. Ρικέ για τη θέση του Συμβουλίου. Η πρόταση που ενεκρίθη από την Κοροπέα την προηγούμενη Παρασκευή και η οποία μάλλον θα είναι τελική, θα οδηγήσει σε περικοπές στις μεταφορές, ιδίως για την ΣΕΣΑ, για την ΙΝΕΑ και κάποιες μικρές περικοπές για τους άλλους φορείς. Εμείς θα χαιρόμαστε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίξει το σχέδιο πρόταση τη Κομισιόν για τι πιστώσεις πληρωμών. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Μασιμιλιάνο Σαλίνη ω συζητητή για να κλείσουμε. Ευχαριστώ όλου του και όλου του συζητητέ για τι ε, παρατηρήσει του. Ακριβώς προχωρήσαμε σε αυτό το κείμενο, ε, όχι μόνο κατά του τύπου, αλλά κατά την ουσία μια συνεργασία. Τώρα ξεκινάω την τελευταία ε, παρέμβαση της Κομισιού Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ένα στοιχείο που απλό, πάρα πολύ βασικό, ότι το ΕΦΣΙ πρόκειται να βοηθήσει με τις ε, εγγύσεις, για πολλές εγγύσεις. Από την άλλη μεριά όμως ε, είναι έτσι φτιαγμένο το ΕΦΣΙ που δεν ωφελεί κάποιο είδους έργα, κάποιο είδου επενδύσεις που είναι μακροχρόνιες και περίπλοκες ας πούμε το ΣΕΦ δεν πρόκειται να καλυφθεί αναγκαστικά από το ΕΦΣΥ και αυτό και αναφέραμε τις εσωτερικές πλωτές οδούς και το σιδηρόδρομο το ΕΦΣΥ πρόκειται να χρηματοδοτήσει ακριβώς ε, κάποιες, κάποιες άλλες, μεταφορές και όχι αυτές που ακριβώς αφορούν κάποιες διαδικασίες μακροχρόνιε. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επενδύσεις οι πιο κρίσιμες προς ώστε να επιτρέψουμε στην ανάπτυξη. Όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση, ε, αυτό είναι που ονομάζουμε ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για τροπολογίες 22 Ιουλίου την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Και η ψηφοφορία θα ακολουθήσει στην Επιτροπή μας στις 31 Αυγούστου που είναι η Δευτέρα μετά τις διακοπές και 28 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης και πρωτού πω οτιδήποτε άλλο θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ, να καλωσορίσω και τον Brian Simpson που είναι δίπλα στην παλιά του θέση είναι αυτός ο οποίος έχει προεδρεύσει την Επιτροπή αυτή στο παρελθόν και έχει λειτουργήσει και ως εισηγητής και ως ε, εισηγητής και χαιρόμαστε που μπορούμε να προσκαλέσουμε τον Ευρωπαίο συντονιστή για τα θέματα αυτά. Ξέρεις πολύ καλά τα κόλπα, ξέρεις να είσαι και σύντομος, έχεις μάθει στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε την ευκαιρία να σε ακούσουμε. Δίνουμε το λόγο λοιπόν στον Brian Simpson. Well, it's a bit strange, I have to say. Λίγο με ξενίζει που πάω μια θέση προς τα δεξιά τώρα που ξαναήρθα στην <laughs> Επιτροπή. Μάικλ, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία σήμερα να μιλήσω για του αυτοκινητοδρόμους, θάλασσες. 505 εκατομμύρια περίπου ε, ζουν στην Ευρώπη σε μια μεγάλη επιφάνεια και άρα ε, από πλευρά μεταφορών για να έχουμε συνοχή και κατάλληλη πρόσβαση στις αγορές και στο εμπόριο χρειάζονται σοβαρές προσπάθειες στον τομέα των μεταφορών. Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες ε, φτιάξαμε τα TEN-T's διότι, τα ΔΕΔ δηλαδή, διότι θα πρέπει να είμαστε πανευρωπαϊκοί και όχι εθνικοί. Μιχάλη, νομίζω ε, σύμφωνες μαζί μου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες γραμμές έχουν εκείνα και ε, να σχεδιάσουμε την επόμενη δεκαετία τα πλαίσια των ΔΕΔ. Τα εθνικά δίκτυα θα πρέπει να λειτουργούν, να είναι διαλειτουργικά. Αυτή είναι η ουσία των ΔΕΔ. Και παρότι ε, στις χερσαίες μεταφορές εξυπηρετούνται περίπου το 60% των αναγκών της εσωτερικής αγοράς, ε, παρόλα αυτά δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι το 40% και ε, χρειάζονται, ουδάλλως έχουμε ε, συμφορές, οικονομικές απώλειες ε, και επιζήμιο αντίκτυπο για το περιβάλλον. Η θαλάσσια σιδηροδρόμο, η, ε, σιδηρο, η θαλάσσια αυτοκινητόδρομη, συγγνώμη, ε, αντιστοιχεί στο θαλάσσιο κομμάτι των ΒΕΔ. Γιατί είναι σημαντική η θαλάσσια αυτοκινητόδρομη, διότι είμαστε Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα των μεταφορών που γίνεται διαθαλάσσι περίπου το 90% και το 40% των εσωτερικών συναλλαγών γίνεται θαλασσίως και 75% επίσης των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών και αυτά γίνονται μέσω ε, θαλασσίων οδών η κατάσταση πως έχει. Έχουμε το, το, τη διόρυγα του ΣΟΕΣ που για να ενωθούμε με την Ασία και με την Ινδία έχουμε τη Μεσόγειο, έχουμε τον Ατλαντικό και το Παναμά, ε, τον ε, Εύξηνο Πόντο και την Πορια Θάλασσα. Ε, την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά εμπορικέ συναλλαγέ ε, με την Ασία και φυσικά αναπτύχθηκαν αντίστοιχα και οι υποδομέ. Ε, κάτω από το 30% των συναλλαγέ μα με τη Δυτική Αφρική και έτσι έχουν συγκεντρωθεί όλα στη διόρυγα του Σουέζε και στη Μεσόγειο και λόγω της οικονομίας κλίματος έχουμε το Ρότερνταμ, το Αμβούργο και τα λιμάνια στο στο κανάλι της Μάχης και εκεί πέρα έχουν συγκεντρωθεί ε, όλες οι εμπορικές συναλλαγές ε, τώρα. Ε, έχουμε το πανομέ για τις οικονομικές τους συναλλαγές με τις ΙΠΑ και ο Ατλαντικός θα χρησιμοποιηθεί τώρα πλέον και τα πλαίσια των αυξημένων εμπορικών συναλλαγών αν εγκριθεί η συμφωνία ε, TTIP. Έχουμε την συνολική υλικοτεχνική αλυσίδα που πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνοχή, όχι μόνο για να καλύψουμε τις τωρινέ ανάγκες, αλλά και για την αύξηση αυτών των αναγκών και χρειαζόμαστε και ποιότητα και ποσότητα στο διατλαντικό εμπόριο. Αν τα καταφέρουμε, θα αλλάξουμε το εμπορικό μας μοντέλο αναγκαστικά, διότι ε, ε, θα χρειαστούν ναι, πολλές και διαφορετικές λύσεις, ούτως ώστε να αποφύγουμε τις ε, τωρινές ε, συμφορήσεις και τα λάθη του παρελθόντος. Ε, ανάμεσα στην ακτή της Ευρώπης ε, και τον ΙΠΑ δεν θα έχουμε οδικές μεταφορές, δεν θα έχουμε φορτηγά πλέον, θα είναι μόνο πλοία που θα πλέουν στον ωκεανό. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε την Ατλαντική ακτή ούτω ώστε γρήγορα να μπορέσουν να ενωθούν ε, τα, με την ενδοχώρα οι μεταφορές που γίνονται μέσω των ε, εμπορευματοφόρων ε, πλοίων. Ε, θα πρέπει λοιπόν επίσης να επιτύχουμε μια ευθυγράμμιση των διατροπικών τρόπων μεταφορών ούτω ώστε να να έχουμε καλύτερη υλικοτεχνική στήριξη για μεγαλύτερη συνοχή και χάρη στις προτεραιότητες ε, των αυτοκινητοδρόμων ε, για την πληροφορική και τα εργαλεία της ε, ψηφιακής οικονομίας θα έχουμε καλύτερη διαχείριση των μεταφορών και θα συνδέουμε όλους τους εμπλεκόμενους χωρίς για κάθε τρόπο μεταφοράς. Αυτά θα τα παρακολουθώ εγώ, γιατί είμαι συντονιστής για τους αυτοκινητοδρόμους τη θάλασσα. Μπορεί να με ρωτήσει κάποιο, μα τι είναι αυτή η αυτοκινητόδρομη. Λοιπόν, ο στόχος συνολικά είναι να έχουμε ένα διευρωπαϊκό δίκτυο θαλασσίων αυτοκινητοδρόμων για τη μεταφορά εμπορευμάτων με τρόπο βιώσιμο και αξιόπιστο, ενοποιώντας δηλαδή τις, θαλάσσιες, τις υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών με μια ενιαία ε, υλικοτεχνική αλυσίδα και έχοντας μια επισκόπηση των μεταφορών. Ε, Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ε, νέε προτεραιότητε ε, στον τομέα των μεταφορών γιατί πέρα από τον δρόμο έχουμε τι συμφορίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι οδικέ μεταφορέ και χρειαζόμαστε πιο βιώσιμού τρόπου μεταφορέ έτσι τι τι αυξάνοντα αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και βελτιώνοντα την πρόσβαση στι περιφέρειε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρω ότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κάποια μέλη της Επιτροπής σας. Εγώ έχω ορίσει τρεις προτεραιότητες ε, όταν δηλαδή ανέλαβα αυτό το ρόλο του συντονιστή για τους ε, αυτοκινητοδρόμους. Ε, περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος, ε, χρήση εναλλακτικών καυσίμων, δύο, ενοποίηση των θελασσίων μεταφορά στην ε, ε, τεχνική αλυσίδα για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν όλοι και στη συνέχεια διαχείριση της ασφάλειας της θάλασσα και ανθρώπινη διάσταση ε, με τα ατυχήματα που έχουν συμβεί θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αυτό ως τρίτη προτεραιότητα. Ο συνολικός μας στόχος ε, είναι να εξυπηρετήσουμε το εμπόριο και να ενώσουμε τα λιμάνια με την ενδοχώρα, να ενώσουμε τα λιμάνια μεταξύ τους και τα λιμάνια με τους διαδρόμους. Τους διαδρόμους με τις τρίτες υπερπόντιες χώρες, ε, είπαμε Μεσόγειος, Εύξηνος πόντου Ατλαντικός ε, και να ενώσουμε την ενδοχώρα μας με τις τρίτες της χώρε. Για τον πρώτο ε, στόχο, για τις προτάσεις ΣΕΦΚΟ, ε, είχαμε 33 εκατομμύρια για τη συνοχή και 630 από το ΣΕΦ. Για τη χρηματοδότηση εγκρίναμε ε, τις προτάσεις για 283 εκατομμύρια και συνολικέ επενδύσει 741 εκατομμύριων. Αυτά και για τα δύο, και για το ΣΕΦ ε, και για το ΣΕΦ. Έχουμε 20 προγράμματα για το περιβάλλον ε, με επενδύσεις 392 εκατομμύριων ευρώ και 147 εκατομμύρια είναι η, η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ελληνικό το υγροποιημένο ε, αέριο έχουμε 6 δράσεις 676 εκατομμύρια σε επιδοτήσεις ε, και χρειαζόμαστε επενδύσεις σε 75 εκατομμυρίων. Ε, για την υλικοτεχνική αλυσίδα και την οποία των μεταφορών έχουμε 5 προγράμματα με 265 εκατομμύρια επενδύσεις. Τα 98 εκατομμύρια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαχείριση της θαλάσσιας ασφάλειας ε, και ο ανθρώπινος παράγοντας, εκεί έχουμε τέσσερα προγράμματα, 82 ε, προγράμματα, 82 ε, εκατομμύρια είναι επενδύσεις και τα 36 από αυτά είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει στο μέλλον. Ε, χρειαζόμαστε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης και θα το λάβετε τον Ιούνιο. ζητώ συγγνώμη, εννοούσα μέχρι το 2021 και ε, μία μελέτη που έχει ξεκινήσει τώρα και θα σας ε, δείξει τους ενδιάμεσους κόσμους μέχρι το 2017. και ε, την ε, ε, ενδιάμεση, ενδιάμεση αναπρογραμματισμό, αναπρογραμματισμό διότι θα, πρέπει, θα χρειαστούμε περισσότερους εμπλεκόμενους φορείς. Ε, υπήρξε υπερκάλυψη επίσης, ε, να το γνωρίζετε γι' αυτό, διότι από τους αυτοκινητοδρόμους, ε, το πρόγραμμα δηλαδή, το περιορισμένο πρόγραμμα που είχαμε, περάσαμε τώρα σε μια πληθώρα προγραμμάτων, υπήρξε υπερκάλυψη λοιπόν. Θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση λοιπόν προς την Επιτροπή, διότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια Ό,τι μπορέσετε να μας δώσετε ε, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Πώς μπορούμε να έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο για τους ε, αυτοκινητοδρόμους. Βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του ΔΕΔΕ που θα καταθέσουμε ε, στο, θα καταθέσουμε στο Κοινοβούλιο και θα κράτημε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για τους αυτοκινητοδρόμους το 2016, Ιούνιο-Ιούλιο μετά από τις διαβουλεύσεις που είχαμε με ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς και θα σας ακούσουμε και εσάς, ε, θα το χρειαστούμε αυτό, ούτως ώστε να γίνει μία διαβούλευση, όχι με βάση γεωγραφικών κριτηρίων, αλλά με κριτήριο την, το τόπο λειτουργία τους, δηλαδή γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μην ξεχνούμε ότι ε, οι περισσότεροι διάδρομοι είναι κάθετοι. Μόνο ένα είναι οριζόντιο και άρα επειδή είναι κάθετοι αφορούν ω ε, επιτοπλίστων ένα περιορισμένο αριθμό χωρών. Όμω εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση σε ολόκληρη την Ευρώπη και γι' αυτό κρίνω πω είναι σημαντικό ρόλο του συντονιστή των αυτοκινητοδρόμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι από τα 400 ε, λιμάνια, δεν ξέρω εγώ πόσα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουμε, είναι πολύ δύσκολο ο συντονισμό και παρόλα αυτά δεν έχουμε χρηματοδότηση στη διάθεσή μα. Και δυσκολευόμαστε ε, σε επίπεδο κρατών μελών ε, για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχή και όχι μόνο αυτό. Θα σα έλεγα ότι εγώ πάντοτε ήμουν άνθρωπο στον σιδηροδρόμο, το ξέρετε αυτό, και ε, είχα αιμονή με αυτό το ζήτημα. Όχι ότι θα θέλω να πάρω τα χρήματα από τους σιδηροδρόμους και να τα πάω στα λιμάνια. Όχι. Απλώς ε, θέλω να σας πω ότι χρειαζόμαστε την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω την τεχνογνωσία σας. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό δίκτυο ΔΕΔ για τους ε, αυτοκινητοδρόμους της ε, θάλασσας το ώστε να κατακτήσει η θαλάσσια μεταφορά και πάλι ε, τον ωκεανό. Και στην ανάλυση των δεδομένων μεταφορών και την κατάρτιση του, του σχεδιασμού θα μπορέσουν οι θαλάσσιες μεταφορές να έχουν ε, το ρόλο που σας αξίζουν, να μην είναι πλέον... Ε, παράνυφος αλλά Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μπράιν. Ε, Βιν Φαντεκάμπ, όχι. Ποιος άλλο αυτό λόγο πάντως. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Σίψον. Εγώ σας είχα αντιμετωπίσει στο παρελθόν ως ε, αντίπαλο πολιτικό, αλλά με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη εκτίμηση, ιδίω όταν ήσασταν πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Περιμένουμε ό,τι καλύτερο από τον κύριο Σίμψον, γιατί είναι ατόφιος άνθρωπος, είναι άνθρωπος που πάντα ενδιαφέρθηκε για τα θέματα των ε, σιδηροδρόμων, όπως ο τωρινός μας πρόεδρος ασχολείται με τα ποδήλατα και τα υποστηρίζει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ο σημαντικός λοιπόν ε, στόχος είναι να έχουμε μια διατροπικότητα η οποία θα είναι αποτελεσματική και οι αρτηρίες της θάλασσας είναι πολύ σημαντικοί για να μπορέσουν να συνδυάσουν μαζί με τους ιδεοδομικούς άξονες τις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διατροπικό τρόπο. Το Connecting Europe Facilities περιλαμβάνει ως οριζόντες προτεραιότητες του, της αρτηρίας της θάλασσας. Και το σχέδιο που μας έχει παρουσιάσει ο συντοριστής περιλαμβάνει τρεις προτεραιότητες. Καταρχήν, το περιβάλλον να μειωθούν οι ρηπαντικές εκπομπές. Δεύτερον, ενσωμάτωση στην ε, αλυσίδα επιμελητίας των θαλασσίων μεταφορών. Και τρίτον, τεχνικές βελτιώσεις της θαλάσσιες μεταφορές. Η σωστή διαχείριση λοιπόν της ε, θαλάσσιας διακίνησης, η κατάρτιση των πληρωμάτων. Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένα να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ε, πλατφόρμα εθμελτίας και να βοηθήσουμε τη διατροπικότητα, να οδηγήσουμε σε καλύτερη ανταλλαγή και μεταφορά των μεταφορών στην θαλάσσια μετακίνηση και όχι στους αυτοκινητοδρόμους. Αυτό είναι κάτι το οποίο λέμε πάντα. Αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει η πιο αποτελεσματική μεταφορά. Να είναι η πρώτη προτεραιότητα των αρτηριών της θάλασσας. Η διάδρομη των μεταφορικών ε, δικτύων χρειάζονται ένα πρόσθετο διάδρομο που είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι αρτηρίες της θάλασσας. Τελικά πρέπει <clears throat> να δοθούν πόροι στους θαλάσσιους λιμένες της Ευρώπης για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τα αέρια θερμοκηπίου. Έτσι <clears throat> θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Είπατε ότι χρειάζεται τη βοήθειά μα. Χρειαζόμαστε, είπατε, περισσότερα χρήματα. Συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Σίμψον. Γι' αυτό δεσμευόμαστε να δώσουμε την πολιτική μας υποστήριξη για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Οι νέοι αυτοί ε, με της θάλασσας είναι σημαντικοί για να αυξηθεί η διατροπικότητα γιατί χωρίς αυτήν δεν θα υπάρξει σωστή λειτουργία ούτε των συνδρομικών συνδέσεων ούτε των λιμένων Επομένως, εμείς υποστηρίζουμε την πρότασή σας και υποστηρίζουμε ότι πρέπει να διακριτήσουμε και περισσότερους πόρους ώστε όλα αυτά να γίνουν σε πραγματικό χρόνο πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ισμαήλ Ερτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Μπράιαν, και εγώ από τη δική μου πλευρά θέλω σε καλωσορίσω θερμά ε, στις συνέντευξη αυτή που γνωρίζει τόσο καλά για μένα και την ομάδα μου <clears throat> είναι μια πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε που σε υποδεχόμαστε και πάλι και ακούμε και πάλι τη φωνή σου. Μια χαρά σε βλέπω και σου εύχομαι και στο μέλλον κάθε επιτυχία στα καθηκόντά σου. Νομίζω ότι σε έχει βοηθήσει το γεγονό ότι έχει αναλάβει άλλα καθήκοντα από το Κοινοβούλιο. Αγαπητέ Μπράιαν, έχει αναφερθεί σε ένα πολύ σημαντικό θέμα και φυσικά έχει σημαντικά καθήκοντα. Ξέρει ότι την τελευταία θητεία του Κοινοβουλίου είχαμε εργαστεί πάρα πολύ στενά για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις κατευθύνσεις γραμμές των διευρωπαϊκών δικτύων όπου εγώ είχα σταθεί συνεισηγητής πολλές φορές επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για αυτό το ζήτημα, για τη στρατηγική αυτή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα Θέλω να τονίσω ότι είναι μια στρατηγική που είναι μοναδική σε παγκόσμιο κόσμο. Μόνο εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήσαμε αυτά τα δίκτυα με σαφεί στόχου, με σαφή προσέγγιση διαδικτύωση, ώστε να μπορέσουμε να προσποριστούμε μια προστέμενη αξία. Είναι λοιπόν μια λειτουργία που ξεκίνησε στο χρονικό διάστημα 2004-2014, αλλά όπως στην πρώτη αυτή περίοδο δεν χρησιμοποιήθηκαν οι ευκαιρίες που μας παρέχουν οι θάλασσες. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν είχαμε κάνει τίποτα. Και σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτηκε, η Κομισιόν συγγνώμη σκέφτηκε ότι πρέπει να αποστεθούν και οι, οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας. Ξέρω πόσο δύσκολο υπήρξε προηγουμένως τους τριλόγους να πείθουμε το Συμβούλιο και τα κρατημέλη ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια πρωτοβουλία για τους αυτοκινητόδρομους στις θάλασσες. Τώρα όταν ακούει κανείς αυτούς τους ε, δρόμους ότι αφορά μονάχα τις παράκτιες χώρες, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ευρύτερο και πολύ σημαντικό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για τις χώρες που είναι χωρίς έξοδο στη θάλασσα. Αναφέρθηκε σε προτεραιότητες, τις οποίες εγώ συμμεριζόμαι απόλυτα, είναι απαραίτητε η μείωση της ε, εκπομπής ε, διοξίδου του άνθρακος, ενσωμάτωση στην αλυσίδα επιμελητίας, σύνδεση σε διατροπικό επίπεδο, γιατί χωρίς όλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία προσθέμενη αξία και φυσικά υπάρχει και το θέμα της ασφαλείας. Θα ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο. Όταν μιλάμε για τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας, θα πρέπει να σκεφτούμε και την γεωστρατηγική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω αυτής της θέσης, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολύ λίγα πράγματα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις στην ε, Βόρεια Αφρική που είναι οι δικές μας αγορές είναι οι πύρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκεφτείτε το κανάλι του Σουέζ η Αίγυπτος είναι μια χώρα ετέρα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο ρεύμα προσφύγων που έρχεται από την περιοχή αυτή. Και επομένω οι αρτηρίε τη θάλασσα, οι αυτοκινητόδρομοι τη θάλασσα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία απαιτούν μια σωστή πολιτική. Δυστυχώ. Το λέω αυτό με δάκρυα στα μάτια. Η θεματική για την κινητικότητα και τη δημιουργία υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα δευτερεύον. Κρίμα είναι αυτό γιατί δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, για τα μεγάλα ονόματα η κινητικότητα και οι μεταφορές είναι κάτι το οποίο είναι παρακατιανό. Άμα δει κανείς το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό εργασίας της ε, Κομισιόν Juncker μόνο πέντε άρθρα υπάρχουν, πέντε παράγραφοι υπάρχουν για τις μεταφορές που είναι γενικά, γενικολογίε. Αυτοί λοιπόν που έχουν αγωνιστεί εδώ και πολύ καιρό για το θέμα αυτό, όλοι οι εμπειρογνώμονε, θα πρέπει να αγωνιστούμε το θέμα αυτό επιτέλους να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει. Και όταν μιλάμε για τα γεωστρατηγικά θέματα, δεν θέλω να αναφερθώ να κάνω την πανοκρουσία, αλλά άμα δούμε τι γίνεται με άλλες ε, χώρες στον κόσμο. Αν δούμε τι γίνεται στην ε, Λατινική Αμερική, αν βλέπουμε ότι πέρα από το κανάλι του Παναμά και η Γουαταμάλα με την Ικαράγουα ετοιμάζονται να φτιάξουν ένα κανάλι και να συνδέσουν τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά εγχειρήματα και έχουν προβλέψει χρηματοδότηση 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αυτό το νέο κανάλι. Όλα αυτά είναι λοιπόν σημαντικά για μας. Δεν πρέπει εμείς απλώς να τσακωνόμαστε για το TTIP, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ και στο EFSI, το πρόγραμμα Juncker, το πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο υποστηρίζουμε βέβαια έχουμε και τις επιφυλάξεις μας γιατί μας έχει πάρει κονδύλια, θα πρέπει να αγωνιστούμε να εξασφαλίσουμε ότι και οι αρτίδες της θάλασσας θα μπορέσουν να ενσωματωθούν μέσα στο EFSI και να μπορέσουν να τύχουν χρηματοδότησης από τους ιδιωτικούς επενδυτές. Εάν γίνει κάτι τέτοιο μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που ανέφερες προηγουμένως. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Ρόμπερ Ντίλ. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Είναι πολύ ευχαριστώ να σε ξανέχουμε εδώ κοντά μας τώρα υπό τον καινούργιο σου ρόλο και ξαναευχαριστούμε για όλα αυτά τα τόσο ακριβή που μας εξήγησε. Έχω δύο θέματα να επισημάνω. Το πρώτα, όπως είπε κάποιες στιγμές, είναι για τις επενδύσεις, τι, γίνεται με το, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Έχουμε, είπαμε για μια επταετία 450 εκατομμύρια. Αυτό είναι το σύνολο της ε, επένδυσης για τις ε, θαλάσσιες αρτηρίες. Άρα πρόκειται για ευκαιρία ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση του νέου δαμείου και έτσι να κατευθύνουμε ε, στις θαλάσσιες αρτηρίες, στις ιδιωτικές επενδύσεις. Και είπαμε αυτό να γίνεται με χαρακτήρα ουδέτερο. Αυτό είναι ακρογωνίος του προγράμματος του Γιούγκερ. Ακριβώ όπως μας ε, έδειξες ε, στο χάρτη, ε, τι γίνεται, θεωρείς ότι θα πρέπει όμως, να καλυφθούν αυτά τα λιμάνια που ανέφερες ή θα πρέπει να καλύψουμε και άλλα λιμάνια γεωπολιτικά πιο σημαντικά. Κάτι άλλο τώρα αφορά εκείνες τις περιοχές που έχουμε ε, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βελτική Θάλασσα, εκεί που έχουμε τον έλεγχο των εκπομπών. Τι γίνεται με το υγρό φυσικό αέριο και τη μεθανόλη. Υπάρχουν κάποιοι φραγμοί στο να αναπτυχθούν αυτές οι περιοχές επί τη βάση των νέων κανόνων ελέγχου των εκπομπών. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα κρύψουμε επεμβάσεις περισσότερες θαλάσσιες αρτηρίες ή πρόκειται αυτή η έλεγχη να είναι απλά ένας φραγμός. Να σα για του νέου διάβλους, για την καινούργια διόρυγα του Παναμά, για τη διόρυγα του Σουέζ. Το είπαμε εκεί για τον Παναμά, στο Eurolat που είχα πει το Μάρτιο. Είχαν πάρα πολλές φορές επιφυλάξεις. Και από πλευρά Νικαράγουα. Γιατί είχαμε πει ότι πολλές φορές έχουμε ε, το να λειτουργούν αυτά τα προγράμματα και τα έργα σαν μια φούσκα η οποία σκάει και το έργο καταραίει. Επίσης να δούμε τι γίνεται και με τη μεταφορά φορτίων για θαλάσσης. Και δίνω Ευχαριστώ πολύ λέει η Ζήνα Μάισνερ. Είναι τεράστια η χαρά μας να σε δούμε εδώ Μπράιαν και είναι πραγματικά συναρπαστικό να σε βλέπουμε να είσαι ο συντονιστής για τι αρτηρίε τη θάλασσα. Ε, και ξέρουμε βέβαια ότι είσαι άνθρωπο των σιδηροδρόμων. Άρα νομίζω ότι καλά θα τα καταφέρει και, και με τα πλεούμενα. Ε, έχω λοιπόν ε, πολύ ενδιαφέρον να δω πώ θα προχωρήσουν τα πράγματα αυτά. Θυμάμαι το 2009 που εγώ είχα εκφράσει το ενδιαφέρον για τη θαλάσσια πολιτική. Εσύ είπε, βρέγγε τι, είναι, τι μου λε τώρα. Αλλά ενδιαμέσως νομίζω ότι έχει καταλάβει τη σημασία των θαλασσίων δρόμων στην Ευρώπη, ιδίως για χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και μια ολοκληρωμένη μεταφορική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να συμπεριλάβει και τις θαλάσσιες μεταφορές. 90% όπως είπε των μεταφορών γίνεται με τη θαλάσσια οδό. Είναι πολύ καλό αυτό να λειτουργεί καλά γιατί αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρώπη και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα διατηρήσει τη θάλασσα καθαρή με το να μειώσει τις ε, εκπομπές. Όπως είπε και ο Έρτουχ, όλα αυτά έχουν και γεωστρατηγικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την ασφάλεια των θαλασσίων οδών της Ευρώπης και χρειαζόμαστε να έχουμε επίσης και περισσότερα σωστικά μέσα, ιδίως με τους μετανάστες που φτάνουν στις ακτές μας. Επομένως, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα που έχει ξαναλάβει. Έχω ένα ερώτημα τώρα συγκεκριμένο ρωτάω πάντα τους ε, συντονιστές κατά πόσο μπορούν να εξασφαλίσουν καλά το συντονισμό. Γι' αυτό το ερώτημα είναι, εσύ θα συμμετέχεις στη στρατηγική για τις θάλασσες λεκάνες, για την Αδριατική Ιόνια Λεκάνη, για την Βαλτική, για τη Βόρεια Θάλασσα, εκεί λοιπόν που οι όμορες, οι παράκτιες χώρες προσπαθούν να συνδυάσουν τις ενέργειές τους, το ερώτημα μου είναι θα έχεις μια παρουσία ή έχεις κάποιους δικούς ανθρώπους οι οποίοι θα παρακολουθούν αυτές τις στρατηγικές. Αν όχι αυτό πρέπει να αλλάξει. Και επίσης ένα ερώτημα, μήπως υπάρχουν προβλήματα με κάποια συγκεκριμένα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να σε βοηθήσουν περισσότερο στην εργασία σου. Ίσως δεν μπορείς να μας το πεις αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εγώ είμαι πεπισμένη ότι χρειαζόμαστε αυτούς τους ε, αυτοκινητόδρομους, αυτές τις αρτηρίες της θάλασσας Πρέπει όλα τα κράτη μας να εργαστούν για να έχουμε και εναλλακτικέ υποδομές για τις ε, εναλλακτικέ ενέργειες και για τη σύνδεση με την ενδοχώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να ξέρουμε ποιες χώρες θέλουν περισσότερη πειθό ώστε να εργαστούμε για τους ε, βουλευτές και τις κυβερνήσεις τους. Και το επόμενο ερώτημά μου είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο Ρόμπερτ Σίλε για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και αυτό το λέω ότι έρχομαι από τη Βόρεια Γερμανία. Πώς βλέπεις λοιπόν την ε, ανάπτυξη αυτή και ποια είναι η αξία των scrubbers, δηλαδή των φίλτρων για τις εκπομπές. Εγώ πιστεύω ότι ε, εάν δεν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτό το υγροποιημένο φυσικό αέριο, δεν θα προωθήσουμε. Και επίσης, τι έχει επιτευχθεί με τους scrubbers, με τα φίλτρα αυτά, για, σε συνεργασία με την ΕΜΣΑ και άλλους φορείς, οι οποίοι ελέγχουν τα θέματα αυτά για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιούν υγρά φίλτρα για να απορροφούν τις εκπομπές. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Σε ποιο βαθμό παίζουν και οι απομεμακρυσμένες περιοχές ένα ρόλο στους, στις αρτηρίες της θάλασσας. Προφανώς αυτό ενδιαφέρει το την υπηρετική Ευρώπη, αλλά τα νησιά μας έχουν πάντα προβλήματα με την πρόσβαση. Θα, σε ποιο βαθμό λοιπόν οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας καλύπτουν και τις ανάγκες των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών. Ευχαριστώ, Εμάγια Κίλονεν. Κύριε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρεμ που ήρθες. Την περασμένη φορά που σε είδα, ήσουν πρόεδρος και εγώ είχα μακριά μαλλιά. Τώρα κουρεύτηκα και έγινα και βουλευτής. θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα που σχετίζονται με τις βόρειες σκανδιναβικές χώρες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, για τη σύνδεση ανάμεσα στο ΟΜΕΟ και τη ΒΑΖΑ σύνδεση δηλαδή, της με τη Σουηδία ε, προβλέπεται χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως ε, για τα ε, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Θα μας ενδιαφέρει να μάθουμε. Επίσης, τι πιστεύεις ε, για τα, τα όρια για το θείο. Πώς επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα των βορείων διαδρόμων. Θα υπάρξει αυστηρή συμμόρφωση και επίση το, το των θαλασσίων μεταφορών θα υπάρξουν μεταφορέ δικαιωμάτων εκπομπών σε σχέση με τι οδικέ μεταφορέ με φορτηγά, παραδείγματο χάρη. Ναι, και μία τρίτη ερώτηση. Στα πλαίσια των ε, ε θαλασσίων αυτοκινητοδρόμων, γενικότερα έχει τεθεί το ζήτημα των μεταφορών ανάμεσα στους διαφόρους διαδρόμους. Ο Βέρνερ Κούν. Και εγώ θέλω να προσθέσω τη δική μου χαρά για την παρουσία σου εδώ, Μπράιαν. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ε, περίοδο με ένα συγκεκριμένο θέμα που θυμάσαι ίσως From Road to Sea, από το δρόμο στη θάλασσα. Η αυτοκινητόδρομοι λοιπόν της θάλασσας είναι η συνέχεια, η λογική συνέχεια μιας πολιτικής για τις οδικές μεταφορές. <clears throat> Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κατηγοριοποίηση σε κεντρικούς ε, λιμένες, το λιμένο του Βορρά και του Νότου και είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ένα δίκτυο αξώνων χερσαίων που να συνδέει αυτούς τους ε, λιμένες. Η αυτοκινητόδομη της ε, θάλασσας έχει παραμείνει άξονα των, ε, διευρωπαϊκών δικτύων χάρη στην δική μας επιτροπή. Στην αρχή δεν φαινόταν πάρα πολύ σαφές ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει δεκτοί οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας ως διευρωπαϊκά δίκτυα ώστε να χρηματοδοτηθούν καταλήλως. Ήταν πολύ σημαντικό βέβαια ότι μπορέσαμε εμείς με, τις, ε, με τους μεγάλους αυτούς οικονομικούς χώρους της ε, Βόρειας Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία και επαφή σε ό,τι αφορά το εμπόριο των μέσω εμπορευματοκιβωτίων. Έχουμε λοιπόν μεγάλα λιμάνια όπως το Ρότερνταμ, το Αμβούργο που έρχονται σε επαφή με την Βόρεια Αμερική και με τις ε, με του, τα πλοία που έχουν 14 ή 21.000 εμπορευματοκιβώτια ισοδύναμα, αυτά έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο πλέον και πρέπει να είναι τροφοδοτικού χαρακτήρα. Να, να βοηθούν να ε, καλύπτουν τα, να τροφοδοτούν τα μεγάλα πλοία με εμπορευματοκιβώτια και θα χρειαστούν και περισσότερες επενδύσεις τους λιμένες ώστε να μπορεί να γίνεται μια καλύτερη κατανομή των φορτίων και να μπορούν να μετακυλίονται σε περαιτέρω μέσα μεταφοράς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά πρέπει να διατηρήσουμε και τη στατική μας θέση. Ξέρουμε ότι αυτοί οι Κινέζοι έχουν πάρει ένα μερίδιο της διαχείρισης του καναλιού του Σουέζ. Τώρα με τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα έχουν πατήσει και το πόδι του στον Πειραιά. Όλα αυτά είναι κρίσιμες υποδομές είναι απαραίτητο λοιπόν η Γερμανική Ένωση να διατηρήσει τη θέση της σε αυτά τα λιμάνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και το θέμα της ειδική ε, χρήσης ενεργειακών πόρων στην θάλασσα ξέρουμε ότι πιο αποτελεσματική είναι η χρήση της ενέργειας της μεταφορές στη θάλασσα από ότι στον, ε, στην ξηρά. Όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με εκπομπέ λοιπόν διοξιδίου του άνθρακο και το ETS είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά να παίξει και κάποιο ρόλο φυσικό αέριο και να βρούμε ένα καλό τρόπο να υπάρξει υποδομή για να διανέμεται το ε, φυσικό αυτό αέριο ως καύσιμο για τα πλοία και για τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας και επίσης θα πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξη για τις βραχίες θαλάσσιες μεταφορές γιατί αυτές οι μεταφορές μας δίνουν μια μεγάλη ασφάλεια Θυμηθείτε τι είναι με το κανάλι ε, από τη Βόρεια Θάλασσα στην Βαλτική και την ε, χρήση του Γκαλιλαίου ως συστήματος πλοήγησης που μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια στη θάλασσα. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία καλύτερης ε, ε παρακολούθησης. Αναφέρθηκε στο Βόσπορο τη διέλευση του Βοσπόρου που είναι η σύνδεση από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Δεν μπορούμε πια να ελέγξουμε το κόστος αυτών των μεταφορών γιατί υπάρχει το πρόβλημα της περιεκτικότητας σε θείο. Στα κάσμα των πλοίων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία των scrubber, των φίλτρων λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή με τις τιμές του πετρελαίου δεν νοιάζονται οι εφοπλιστές πια να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες scrubber ή φυσικό αεριγροποιημένα. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει και εσύ, Brian. Η Τερέζα Γρίφιν τώρα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι υπέροχο το ότι βρίσκεσαι εδώ, Μπράιαν. Ε, Ξέρουμε ότι δεν είσαι πια ευρωβουλευτή, αλλά γνωρίζουμε ότι όπω και τότε που είχε πετύχει τόσο πολλά στην Δυτική Αγγλία, είσαι και τώρα πάρα πολύ ε, ενεργός και είπαμε ότι ε, ε, γι' αυτό τον, πρέπει να δούμε πού, πού έχουν πέσει οι μεταφορές, πού υπάρχει κάποια παραγμή, πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας που εχουν πεσει οι μεταφορες που υπαρχει καποια παραγμη πως θα δημιουργησουμε θεσεις εργασιας που θελουμε στο θεματολογιό μας να το εντάξουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εσύ προσπαθείς να βοηθήσεις σε εκεί στη βορειοδυτική Αγγλία τον λιμένα του Λίβερπουλ και κατά αυτόν τον τρόπο πώς θα έχουμε με αυτές τις αρτηρίες, της θαλάσσιες, πώς θα τονώσουμε την Προεδρική Αγγλία και το Λιβερπούλ. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα ε, έχουμε τα προτύπα που ξέρουμε για όλου του εργαζόμενου και πώ θα έχουμε κάποιες μαθητείες ε, και κάποια στάζ για του εργαζόμενου εκεί, τι θα γίνει με τις γυναίκες ναυτικού είναι μόνο 2% και 21% ε, των συνολικά εργαζομένων στις μεταφορές. Άρα εδώ ε, έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Δεν λέω ότι όλα αυτά εσύ θα πρέπει να τα λύσει. Απλώ πε μα πώ μπορεί να συμβάλλει. Δεν Φαντεκάμπλε, πρόεδρο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαι ο μόνος εδώ στην Επιτροπή μας που δεν έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής μας επί Προεδρίας Σίμψον. Αλλά όμω ε, είχα συντάξει ε, όταν ήμασταν μαζί στην ΙΜΚΟ μια έκθεση. Πάντως πολλά αλλάξαν από τότε, Μπράιαν, μάλλον τώρα χειρότερα τα πράγματα. Έχω να σου υποβάλω τις εξή ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά την ανακοίνωση συγγνώμη την επικοινωνία. Τι κάνει το επιτελείο σα ε, κύριε Σίμψον σχετικά με αυτό. Είπαμε ότι εμείς ξέρουμε τι είναι δράση αρτηρίας, αλλά ξέρει ο κόσμος στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να κατευθυνθεί μια προσπάθεια επικοινωνία σχετικά με τις θαλάσσιες αρτηρίες. Δεύτερον, μας εξήγησατε πώς έχει κατάσταση των πραγμάτων σήμερα, αλλά δεν κατάλαβα κάτι. Τι θα κάνετε μεταξύ 2014 και 2020, εδώ λέμε για κάποια έργα μεταξύ 2007 και 2013 σε αυτό το φάκελο. Θα έχουμε αναχείραση. Επομένω, τι θα γίνει μεταξύ του 2014 και του 2020. Άλλο. Έχουμε καλή συνεργασία ως συντονιστές, αλλά ίσως καμιά φορά είναι δημιουργικό το να υπάρχουν κάποιες ε, αντιθέσεις. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Μόνο με γλύκες και ευγένειες δεν βγαίνει τίποτα. Τέλος πάντων για τον IMO τώρα. Φυσικά και έχουμε πάρα πολλά θέματα που καλύπτονται από τον IMO. Συνεργάζεσαι με τον ΑΕΜΟ ή θεωρείς ότι δεν είναι αρμοδιότητά Τώρα επίσης όσον αφορά την νομοθεσία για τους λιμένες. Μας έχει απασχολήσει αρκετά. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ λιμένων. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Τι λες γι' αυτό. Yeah, it's Keith Taylor. Oh, Keith Taylor. Well, hello, Brian. Γεια σου, Brian. Nice to see you again. You're looking very well. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, μια χαρά μου φαίνεται. Δύο απλά ερωτήματα έχω μόνο. Ίσως το μπορούσες να πεις κάποια πράγματα. Με ποιο τρόπο οι αυτοκινητόδρομοι θα βελτιστοποιήσουν το δυναμικό του short shipping. Έχεις παραδείγματα βελτίστων πρακτικών. Δεύτερη ερώτηση. Η διασυνοριακή ενοποίηση και η συνεργασία διαφορετικών ε, λιμένων με ποιον τρόπο μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δρόμων. Αν μπορείς, μου ε, ξαναλες το, το δεύτερο, η δεύτερη ερώτησή σου ποια ήταν, έλεγα πώς η διασυνοριακή ε, ενοποίηση και συνεργασία λιμένων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους αυτοκινητοδρόμους. Για να δούμε τι πώς να πεις για το... Ο Γιώργος Μπαχ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες, ε, Μπράιν, και από τη δική μου πλευρά. Το οι χαιρετισμοί από όλου δείχνουν πόσο δημοφιλή είσαι στην Επιτροπή μας. Ελέγχθησαν πολλά για τη χρηματοδότηση υποδομών, της ε, αλυσίδα επιμελτίας. Αυτό το σημείο που με ενδιαφέρει εμένα ήταν το τρίτο σημείο το οποίο ανέφερες, η διαχείριση τη κίνηση και το ανθρώπινο στοιχείο. Ξέρουμε ότι στο ορατό μέλλον δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ε, πληρώματα ευρωπαϊκά στα πλοία μας ε, και σε άλλες μορφές μεταφορών. Στη θάλασσα όμως χρειαζόμαστε ε, ανθρώπους από τις Φιλιππίνες και πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για την εκπαίδευση του ανθρώπινου στοιχείου που αυτή τη στιγμή παίρνουμε από τρίτες χώρες και επανδρώνει τα πλοία μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, Μπράιον. Ε, για όλους εμάς εδώ από το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι χαιρόμαστε που ήρθε σήμερα. Θα ήθελα να ε, τονίζω αυτό που είπε και ο Ισμαήλ, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η πτυχή της χρηματοδότησης. Τι προβλέπεις για το μέλλον για τα προγράμματα για το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπω ότι αυτά που έχουν τη χρηματοδότηση γέφυρα προχωρούν. Το χρειαζόμαστε αυτό. Για τα μεγαπλοία τι προβλέπεις, ε, ε, έχουμε και την έκθεση του ΟΣΑ για αυτό το είδος ε, πλοίων. Πώς πιστεύεις ότι αυτό θα επηρεάσει τους στόχους των αυτοκινητοδρόμων, κυρίως για τη βιωσιμότητα, διότι από κάποιες πλευρές είναι θετικό, αλλά δημιουργούνται και προβλήματα. Συμφωνώ με αυτά που είπε η Τερέζα για τις ποιοτικέ θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη και χαίρομαι που υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο για την κατάρτιση. Για τα άλλα ζητήματα τι κάνουμε, παραδείγματος χάρη για τους ναυτικούς. Την περασμένη εβδομάδα ψήφισε το Κοινοβούλιο ούτω ώστε να υπάρχουν κατοχυρώμενα ισχυρά συλλογικά δικαιώματα για τους ναυτικούς. Πολύ σημαντικό αυτό. Όμως έχουμε και τις σημαίες ευκαιρίας ε, και ένα αγώνα προ τα κάτω. Αυτό επηρεάζει γενικότερα ε, την ποιότητα των θέσεων εργασία. Οι συνάδελφοι από του σοσιαλιστές και δημοκράτες προσπαθούν το φθινόπωρο να διοργανώσουν ένα σεμινάριο για την πρόοδο, για τα κοινωνικά ζητήματα και τα συλλογικά δικαιώματα των ε, ναυτικών. Ε, πώς βλέπεις, τι βλέπει για το μέλλον, Ντομινίκ και Ευχαριστώ, Μπράιαν παρότι ε, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία από πολιτική σκοπιά. Εγώ καθόμουν στα αριστερά σου για πέντε χρόνια. Χαίρομαι ε, που σε βλέπω σήμερα. Να προσπαθήσω να εξηγήσω την ερώτηση που έχω. Σταμάτησε η πρωτοβουλία Μάρκο Πόλο και αυτή η πρωτοβουλία σχετιζόταν με την ενδοκινοτική θαλάσσια σύνδεση, σύνδεση λιμένων. Και τι γίνεται με τους αυτοκινητοδρόμους υπάρχουν ε, θέματα υποδομών, δηλαδή να έχουν λυμμένες τις ε, κατάλληλες υποδομές. Ε, και λοιπόν πέρα από το θέμα της ενδοκινητικής ε, σύνδεσης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτές οι γαλάζιες αρτηρίες ε, είναι η προέκταση με τα ίδια μέσα και τα ίδια πλοία του που χρησιμοποιούνται για τις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές ε, προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρειάζεται ειδικό εξοπλισμός για, του, για τις θαλάσσιες αρτηρίες και αν ναι, ε, τι δυνατότητες υπάρχουν διότι το ΣΕΦ στα πλαίσια των ΔΕΒ δεν ε, προβλέπει για τα πλοία, ε, πόρους ε, για τον εξοπλισμό εκτός ε, από τις εκπομπές των σκράμπες και κάποια, κάποιους πόρους για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται. Αλλά κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα είναι για τους λιμένες. Σε ξαναρωτώ λοιπόν, μπορούμε να προβλέψουμε για το short shipping συγκεκριμένα πλοία, δηλαδή κατάλληλα εξοπλισμένα πλοία. Ευχαριστούμε, Τζέκη Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό να που ξαναβλέπω τον Brian εδώ. Είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ. Ήταν πάντα με στην καρδιά μας. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι μέσα στις αρμοδιότητες σας, αλλά ίσως θα πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί σίγουρα ε, έχουμε περάσει πολύ χρόνο να πηγαίνουμε σε διάφορα λιμάνια την Ευρώπη και αυτό το οποίο ήρθε στην προσοχή μας είναι ότι θυμάσαι ίσως όταν ήμασταν εδώ ότι είχαμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος η DG Trans είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό είναι η οδηγία για το θείο το θιάφι δηλαδή όχι το θείο γιατί αυτό είχε εισαχθεί στη Βόρεια θάλασσα αλλά όχι στην ε, Μεσόγειο και πολλές εταιρείες έχουν δαπανίσει πολλά χρήματα για να πάρουν όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να μειώσουν τις εκπομπές. Αλλά υπάρχει και μια άλλη οδηγία που είναι η οδηγία του καθαρού νερού που αντιμετωπίζει η, Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μια σύγκρουση, μπράιαν και δεν ξέρω αν μπορείς να συμφιλιώσεις τις δυο αυτές τις πληγές Έχουμε την ε, τον τομέα τον αφιλιακό που κάνει μεγάλη προσπάθεια να συμμορφώνεται με την οδηγία για το θείο και πηγαίνει τώρα σε διάφορα λιμάνια που λένε ότι σύμφωνα με την δομική νομοθεσία δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτόν τον εξοπλισμό για να, στον ανεφοδιασμό με τα, τα καύσιμα. Και όταν μιλήσετε στην Γενική Διεύθυνση για το περιβάλλον λένε ότι το καθαρό νερό είναι καλύτερο από το καθαρό θείο, ότι έχει προτεραιότητα από τα καθαρά καύσιμα καλύτερα. Αυτό το οποίο κάναμε τώρα είναι πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά λεφτά με καλή πίστη έχουν κάνει αυτό το οποίο τους λέμε και τώρα τους αφήνουν στα κρύα του θείου γιατί κανείς δεν έχει πάρει μια απόφαση για το πώς θα μπορέσουν να είναι καθαρά και τα νερά και ο θείος. Το έθεσα το θέμα αυτό λοιπόν με την DG Move εξ ονόματο των αυτιλιακών αυτών κύκλων και προσπαθούν να το εξετάσουν αλλά και η DG Περιβάλλον είναι τμήμα τη Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να κάνει κάτι γιατί δεν υποχωρούν καθόλου. Μήπω μπορώ να σου δώσω αυτό δεν περιμένω να μου δώσετε μια απάντηση, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει σύγκρουση των τοπικών κανονισμών σε ορισμένα λιμάνια με εναντί των οδηγιών μα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όταν θέλουμε να έχουμε μια ατζέντα οικονομική μεγέθυνση και έχουμε τόσο σημαντικό ναυτιλιακό τομέα σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ζητήσω αν οι καλέ σου υπηρεσίε μπορούν να οδηγήσουν σε μια βελτίωση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ και τώρα έβαλα και εγώ τον εαυτό μου τελευταίο στον κατάλογο μιλητών, όπως έκανες και εσύ τα παλιά καλά χρόνια. Το ερώτημα είναι τώρα το εξής που θέλω να σου θέσω. Είναι φανερό ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της, ε, των θαλασσίων θεμάτων και του Προέδρου κάθε επιτροπής. Ο τελευταίος ήταν ο Πάολο Κώστα, ο οποίος ήταν ε, και ο επικεφαλής του ο πρόεδρος του λιμένος της Βενετίας. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει και με ψένα μια σύνδεση. Το θέμα λοιπόν είναι αν κάποια κράτη συνδυάζουν τις προσπάθειές τους και έχουν ένα κοινό προϊόν. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Δεν δίνουμε αρκετή βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη δική μου χώρα η γερμανική κυβέρνηση θέλει να έχει μια γερμανική πολιτική λιμένων. Και οπότε υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ των ομοσπονδιακών κρατηδίων στην ε, Γερμανία, διότι έχουν διαφορετικές απόψεις. Το Wilhelmshaven, χάρη είναι ένα κακό παράδειγμα. Δεν μπορούν τα πλοία από το Wilhelmshaven να πάνε στο, δεν να πάνε στο Αμβούργο. Τώρα έχει τελειώσει το λιμάνι, αλλά είπε το το Αμβούργο, όχι να φτιάξετε να διευρύνετε τον Έλβα ώστε να έρχονται τα πλοία στο Αμβούργο και όχι στο Βίλεμς Χάβεν. Επομένως υπάρχουν συνέχεια αυτές τις συγκρούσεις αρμοδιοτήτων ή διευρύνουν τους λιμένες ή φτιάχνουν νέους λιμένες. Αλλά μα γίνεται κάτι τέτοιο με το να υπάρχει χρήμα για την διεύρυνση του ΕΛΒΑ, αυτό κατεδαπάνει σε ευρωπαϊκό χρήμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι σπατάλι γιατί δεν πετύχαμε τίποτα και συμφωνώ με την Γεζίνη για το θέμα αυτό. Και το δεύτερο είναι το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία. Σημαντικό λοιπόν για μένα είναι η ναυσιπλοεία στην ανοιχτή θάλασσα χρησιμοποιούν το, το πετρέλαιο μπούνκερ που είναι το πετρέλαιο αυτό το οποίο είναι το πιο βαρύ κατάλοιπο της επεξεργασίας του πετρελαίου. Με αυτόν τον τρόπο ε, ε, ε, κάνε εξοικονόμηση λιγάκι, αλλά με τον τρόπο αυτό κατα, καταστρέφουν το περιβάλλον, ενώ αν το κάνουν αυτό με, με φίλτρα, τότε θα κοστίσει λίγο περισσότερο, αλλά το συνολικό κόστος είναι πολύ μικρότερο. Πόσο καιρό λοιπόν θα συνεχίσει αυτό το παιχνίδι και τι θα κάνεις για αυτές τις παρακάμψεις της νομοθεσίας. Και τώρα Brian, πολλές ερωτήσεις, αλλά έχεις το λόγο. Simpson. Με σειρά να απαντήσω. Όταν ξεκινήσαμε με τα θέματα αυτά τα υλικοτεχνικά, για να δούμε τι γίνεται σε ποια είναι η σχέση τέλο πάντων αρτηριών και των λοιπών διαδρόμων πρώτα πρώτα, ε, να ξεδιαλύνουμε το κατά πού πήγαινε η ροή της κυκλοφορίας. Οπότε είπαμε να συνδέσουμε τον σιδηρόδρομο με το λιμάνι σε συγκεκριμένες περιοχές και σημεία. Γιατί είπαμε ότι δεν ωφελεί να έχουμε ένα υπέροχο λιμάνι, υποδομή και όλα κομπλέ, εάν, εάν το φορτηγό τρένο κολλήσει σε ένα σημείο συμφόρησης 5 μίλια από το λιμάνι ή 5 μίλια από το λιμάνι. Ε, πιο μακριά δηλαδή, πιο κοντά. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει αυτό αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα να εξεταστούν και να δούμε το πώς τα φορτηγά τρένα θα λειτουργούν καλύτερα. Διαβούλευση, είπαμε ότι είναι βασικό για να εξετάσουμε τα θέματα τα λίγο τεχνικά. Και είπαμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η διαδρομή εργοστάσιο μέχρι τον πελάτη. Εδώ να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική απρόσκοπη λειτουργία για το περιβάλλον Σύμφωνα, μπορεί κανείς να την κουβέντα αυτή να τη συνεχίσει επάρχον. Όμως, είπαμε ότι έχουν αυτή την περιοχή την ελεγχόμενη ε, στη Βαλτική. και αυτά τα μέτρα τα έχει επιβάλλει ο ΑΕΜΟ. Ζήτησαν παρατάσεις, δεν τους δόθηκαν, οπότε ε, είπαμε ότι τώρα έχουμε εκεί την ε, λιγότερη χρήση ε, καυσίμων τα οποία περιέχουν θείο. και τους είπαμε ότι, ότι τελικά έτσι θα γίνει, θα πιάσει τόπο αυτή η πολιτική. Υπάρχει τώρα η υποδομή, έχουν γίνει μετατροπές στα σκάφη και τους είπαμε θα τους βοηθήσουμε. Να τι κάναμε. Κατάλαβα ότι πέρασε το μήνυμα ότι δύο χρημάτων. Και δεν γνωρίζετε αν λεφτά, αλλά μας ενδιαφέρει το δικό μας project, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει, ε, γιατί είπαμε να φέρουμε μια καινοτομία, αλλά ήδη ε, καθυστερήσαμε τελικά σε σχέση με τη λειτουργία των διαδρόμων. Το θέμα είναι βέβαια το πώς κανείς θα προτάξει καλύτερα τα επιχειρηματότητα. Περισσότερα δηλαδή τρένα, περισσότερες αρτηρίες, θαλάσσιες κλπ. Δεν το έχω κολλήσει αυτό το σημείο, αλλά είπαμε ότι έχουμε καλά έργα και προγράμματα τα οποία απορρίπτονται. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Και δεν λέμε τώρα να μεγαλώσει το καρβέλι, αλλά θέλουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από το δεδομένο καρβέλι, δεδομένη πίτα. Είπατε ειδικά τα όσα ισχύουν όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και είπαμε ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της ε, πολιτικές μας μεταφορών. Είπαμε να εμπλακούν όλοι και νομίζω ότι ξεκίνησε η διαδρομή των διαδρομών δικτύων το 1991, οπότε και τότε κάθε ευρωβουλευτής ήθελε να ωφεληθεί το, το αγαπημένο του πρόγραμμα. Άλλος για δισκοτία ή οπουδήποτε. Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει κάποιο να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο, να συνεργαστεί με τα κρατή μέλη, να δει τι χρειάζονται και θα πρέπει μετά να έχει συνέπεια. Και έτσι να πετύχει κάτι. Και νομίζω ότι καλά τα πάμε προς αυτό το μέτωπο. Η είναι πάντως ότι πάντοτε υπήρχαν οι θαλάσσιες αρτήριες αλλά απλώ τώρα το συνειδητοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί υπάρχουν μεγάλα θεματολόγια, αλλά ανακαλύψανε τώρα τι θαλάσσιες αρτηρίε. Όντω το έργο μας το αγνούσαν οι περισσότεροι. Τώρα όμω πιστεύω ότι έχει περάσει το μήνυμα. Τα είπα και στους συντονιστές. Αφήστε πάνω μου τα λιμάνια. Εγώ σας το αναλαμβάνω. Θα βιώσουμε με τα λιμάνια στο δικό σας ε, διάδρομο και με τους πόρους που έχετε διαθέσιμους εσείς και νομίζω ότι αυτό είναι η συνταγή επιτυχίας. Και κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει αναγνώριση όσον αφορά τους λιμένες και τις θαλάσσιες μεταφορές. Τώρα, ε, για τα γεωστρατηγικά, τη, ε, τη, τη, ε, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να μάθουν οι τρίτες χώρες τι πρεσβεύουμε. Η Βόρεια Αφρική, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Μαύρη Θάλασσα. Και για τα ευρωπαϊκά δίκτυα είδαμε πως ε, ε, είχαμε κάποια project με την Παλαιστίνη ας πούμε, αλλά και με Καναδά, Ισραήλ, ΙΠΑ ε, και οπότε έχουμε τελικά αυτόν τον νέο διάδρομο, σύνδεση με Ιταλία και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο σιδηρόδρομος προς την υπόλοιπη Ευρώπη Οπότε είχαμε πει ότι θέλουμε παλαιστινιακά αυθεντικά προϊόντα, όχι παλαιστινιακά τα οποία έχουν ε, παραχθεί στα κατεχόμενα από το Ισραήλ. Υπάρχουν, υπάρχουν κάποια έργα και σχέδια που προχωράνε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέσουμε και να εμπλέξουμε τις τρίτες χώρες. Δεν μπορεί να έχουμε μία θαλασσία διαδρομή που να έχει μόνο μία άκρη, που να έχει αφετηρία και τέρμα. Και στη μία άκρη αυτής να είναι μια ακρη αυτη να χώρα. χωρα ε, μιλάμε για στρατηγική επένδυση που είναι ένα δις για, σε, σε τρεις δόσεις για τρία χρόνια. και είπαμε ότι είναι επιλέξιμο οποιοδήποτε λιμάνι που καλύπτεται από τα TNT, τα ευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. Να, ας πούμε, το Ροστόκ είναι επιλέξιμο. Στη Σουηδία, στην Φιλανδία, έχουμε, έχουμε εκεί κάποια κοινά λιμάνια, τα οποία και αυτά είναι επιλέξιμα, επομένως ό,τι βρίσκεται στα ευρωπαϊκά δίκτυα μπορεί να καλυφθεί. Βαλτική και εκεί ήταν ε, μια πρόκληση και μας δόθηκε η ευκαιρία κάτι να πετύχουμε. Οπότε και ασχοληθήκαμε εντατικά με τις βαλτικές χώρες όσον αφορά τα, τα, καύσιμα, το, το υγρό, γκροπημένο φυσικό αέριο. να βήματα τα προοδοτική βοηθήσαμε σε κάποια έργα στα πλαίσια των όσων προβλέπουν οι κανόνες που ισχύουν. Για τη διόρρογια του Παναμά. Υπάρχει ίδια. έχουμε 20.000-30.000 τονάζ το οποίο καλύπτεται. τέλο πάντων μονάδες περιεκτών και θα πρέπει αυτό να δούμε τι θα γίνει κι αλλού πώς θα το ρυθμίσουμε γιατί 30.000 ε, τόνοι, τέλος πάντων 30.000 μονάδες περιεκτών είναι δυνατόν να αφορά οποιοδήποτε σημείο. Τι είναι. Και τι δηλαδή. Τώρα για την πολιτική μας. Ο πιο φανατικός είναι αυτός που προσελκύστηκε. Οπότε και εγώ ακριβώ τώρα ε, ασχολούμαι σαν τελώς τα θέματα της πολιτικής της θάλασσας γιατί έχουμε 90% που περνάει από τη θάλασσα αλλά θα πρέπει να ασχοληθούν πολύ περισσότερο. Ασχολούμαστε, ασχολούμαστε δυσανάλογα λίγο. Και αυτό γίνεται με θαλάσσιες αρτηρίες. Ότι στην αρχή ήταν δύσκολο να πιστούν οι υπόλοιποι συντονιστές. Πολλοί συνάδελφοι επίστηκαν τελικά αφού του μίλησα δύο φορές. Αυτοί που ήταν στην πρώτη συνάντηση και αυτοί που ήταν στη δεύτερη, εν πάση περιπτώσει δέχτηκαν και τώρα συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι το θετικό. Ασχολούμαστε επίσης και με τους λιμένες των εσωτερικών πλωτών υδάτων. στρατηγικές για τη θάλασσα, ναι, και ε, αυτό το καλύπτουμε. Ναι, φυσικά και έχουν προβλήματα με ένα κρατημέλη, αλλά δεν μπορώ να κατονομάσω τώρα κάποια χώρα. Αλλά υπάρχουν προβλήματα με τις χώρες της συνοχής, γιατί θέλουν να δαπανίσουν όλα τα χρήματα στους σιδηροδρόμους. Και Πρέπει κανεί να τους πείσει περί του αντιθέτου. φυσικό αέριο. Και αυτά ε, τα, τα, σκάφη αυτά, είτε είναι υβριδικά είτε είναι καθαρό ένα σκράμπερς, τα οποία σαρώνουν το βυθό, στην περιφέρεια και όχι μόνο, στις 14 Νευρίου νομίζω έχουμε, όχι στις 20, στις 20 διορθώνει ο κύριος Σίμψον στις Βαλιαρίδες μια σύσκεψη όσον αφορά ε, την, την περιφέρεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα συνδέσουμε αυτές τις, ε, την περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις θαλάσσιες αρτήριες. Στον αφορά το Midway Alignment. Ναι, ναι, και αυτό θέλουμε να το προωθήσουμε. Θα πάω εκεί δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου, οπότε η κυρία Κίλινεν, δεν ξέρω, δηλαδή, το τώρα είπε ότι έχει κόψει τα μαλλιά της και εμένα γίνανε η γκρίζα, οπότε τέλος πάντων κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε. Να το ολοκληρώσουμε τώρα όσον αφορά τη Βόρεια Ευρώπη, τις Βόρειες θάλασσες. Είναι απίστευτο το τι γίνεται εκεί. Το πίστεψα μόνο όταν το είδα. Για παράδειγμα, τι γίνεται το χειμώνα όσον αφορά την ναυσιπλοεία. Τι γίνεται με τα παγωθραυστικά. Βοηθάμε Φινλανδούς, Σουηδούς, τις κοινές του προσπάθειες για τα παγωθραυστικά. Έχουμε και επίσης κάποια φεριμπό, τα οποία και αυτά έχουν ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας για τον πάγο. Μεθανόλη είναι ένα από τα θέματα που αφορούν και τη Βαλτική. Επίσης είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε. Περισσότεροι από ένα το αναφέρατε. Δηλαδή το πώς γίνεται η αστυνόμευση. Και πώς γίνεται τέλος πάντων ο έλεγχος του αν εφαρμόζεται η οδηγία για το θείο. Με έχουμε επομένως ε, ένα πρόγραμμα κοινό ούτως ώστε να συντονίσουμε τις αρχές για να επιβλέψουν την τήρηση της οδηγίας. Η Σουηδία, Φιλανδία, περισσότερο συμμετάσχουν, οι περισσότερο να συμμορφωθούν οι βαλτικές χώρες και να υπάρξει επομένω η συμμόρφωση για το θείο. Χέλμοντ. Κάτι για ε, καταξηράν μεταφορές και την Επιτροπή. Ναι, αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που κάναμε, διορθώσαμε αυτό που θέλαμε. Τώρα επίσης ε, η ναυσιπλοεία σε μικρότερες αποστάσεις ε, και αυτό μας απασχολεί στην Κοπενχάγη είχαμε μια συνάντηση και τα συζητήσαμε τι προβλήματα υπάρχουν, τι χρειάζεται αυτή η ναυσιπλοεία short sea shipping νομίζω ότι είναι κάτι σαν καταλήτης για τις θαλάσσιες αρτηρίες να, να είμαστε ειλικρινείς είναι η ατομομηχανή, είναι ε, πολύ βασικός παράγον, βασικός, βασικό κίνητρο. Οπότε προσπαθούμε να επενδύσουμε και στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Και επενδύουμε και στη χρήση μεθανόλης. Και φυσικά πρέπει να βελτιώσουμε και τις ε, εγκαταστάσεις των λιπέν. Για την Τερέσα. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ανανέωση στους λιμένες της Ευρώπης. Το Λίβερπουλ, η, Βρέστη και άλλα ατλαντικά λιμάνια. Έχω πει πολλές φορές. Το Λίβερπουλ για 40 χρόνια που είναι η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στη λάθος μεριά της χώρας. Τώρα είναι στη σωστή μεριά όμως της χώρας και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε το Wilkenock και το Δουβλίνο είναι και αυτή στην ε, σωστή μεριά. Το εμπόριο είναι πάρα πολύ, το, η, κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Εκπαιδεύουμε όχι μόνο τους ναυτικούς με την παραδοσιακή έννοια, αλλά και ναυτικούς που εκπαιδεύουν άλλους ναυτικούς στα κουραζιερόπλαια για να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις και επικοινωνούμε βέβαια με όποιον θέλει να μας ακούσει. Και η μπροσούρα είναι απλώς ένας ε, οδηγός. Η μελέτη που θα παρουσιάσουμε είναι πολύ ενδιαφέρουσα. That's where the detail will be. Αυτά είναι λοιπόν τα σημαντικά για τα σχέδια τα οποία έχουμε ενώπιον μας. Ε, σας είπα ότι αυτή η μπροσούρα ήταν απλώς ένας ε, ε, οδηγός, αλλά η μελέτη θα έχει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Τι σκέφτομαι τώρα για την οδηγία για τα λιμάνια. Περνάω στην επόμενη ερώτηση. Μα τόσες πολλές ερωτήσεις, παιδάκι μου. Οι βραχίες θαλάσσιες μεταφορές. Ντόβερ καλέ. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ καλή περίπτωση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μιας ε, σύντομης θαλασσίας διαδρομής. Και για τη Βαλτική επίσης. Από το Βάσο στο Ούμιο, πώς τα προφέρνω αυτά τα πράγματα δεν τα καταφέρνω. Διαχείριση της κυκλοφορίας. Ο Τζόρτς το έθεσε το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στον διάβλο της μάχης. Υπάρχει θέμα διαχείρισης της κίνησης και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη Μόνα Λίζα για τη σωστή διαχείριση. Χρηματοδότηση. Τα πλοία μεγαλώνουν. Η αγορά θέλει πιο μεγάλα πλοία. Big is beautiful. Το κόστος του να φέρεις ένα κοντέινερ από την Κίνα στην Ευρώπη είναι πια 200 δολάρια. Αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Από τη Σανγκάη στο Ρότερνταμ 200 δολάρια μονάχα. Από το Ρότερνταμ για να τα πάτε στην Αγγλία μπορεί να κοστίζει περισσότερο. Τα δικαιώματα των ναυτικών μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα θέματα αυτά το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι αυτοί οι ίδιοι ως ανθρώπινα όντα με τα πλοία στα οποία είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν έχουν πρόβλημα. Ακολουθούμε τις διεθνείς συμφωνίες. Ο Μάρκο Πόλο δίνει επιδοτήσεις σε διαδρομές θαλάσσης. εμείς δίνουμε χορηγήσεις σε συγκεκριμένα σχέδια. Ξέρω ότι υπήρξε πρόβλημα με την Ισπανία και τη Γαλλία. Και εγώ τους λέω ότι εγώ είμαι στο Motorways of the Sea, τους θαλάσσιους διαδρόμους και όχι στο Μαρκοπόλο και κάνουμε κάτι που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο και όχι με τις διαδρομές που επιδοτεί το Μαρκοπόλο. Καθαρά νερά. Μίλησε για τους υβριδικούς, τα υβριδικά φίλτρα η Τζάκη. Ναι, τα υποστηρίζουμε στα λιμάνια να υπάρχουν η κατάλληλη, κατάλληλη υποδομή υποδοχής και θέλουμε οι ανοιχτοί, τα ανοιχτά φίλτρα να γίνουν κλειστά φίλτρα που μπαίνουν στο νερό ώστε να μην παραδιαστεί η οδηγία περί των καθαρών νερών. Ε, πρόσφατα συνάντησα τον Παύλο Κώστα. Είναι καλό αυτό το σχέδιο. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να πείσει τα λιμάνια να συμμετάσχουν. Είναι πολύ καλό λοιπόν αυτό το σχέδιο για τα λιμάνια της Βόρειας Αυδιατικής. Το να υπάρξει σύνδεση των λιμένων αυτό πρέπει να είναι μια πρωταρχική προτεραιότητα για όλους μας, για όλα τα κράτη-μέλη. Είχαμε προβλήματα στα κράτη-μέλη και αν με βοηθήσετε σε αυτό θα μου κάνετε μια πολύ μεγάλη χάρη. Θέλω να ξέρω γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό τα σύνορα χωρίς πρόβλημα, αλλά θέλει κανείς να περάσει ένα πλοίο από την Ισπανία στην Μεγάλη Βρετανία πρέπει να περάσει από τελωνιακές διατυπώσεις, λιμενικές διατυπώσεις και όλα αυτά. Δεν φαίνεται να έχει νόημα αυτό. το Αμβούργο και το Βίλιαμ Σχέιφεν. Αχα. Είπαμε για τον Έλβα, για, τη διαπλάτηση, για την ε, διαβάθμιση του Έλβα, αλλά Τους έχω ρωτήσει ήδη για το Κιλ ε, ε, που είναι ακριβώς δίπλα, αλλά ακόμη δεν μου έχουν πει τίποτα. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι ως πρόεδρος δεν θα έχω ποτέ την ευκαιρία να μιλήσω τόσο μακροσκελός όσο εσύ τα κατάφερες σήμερα. Ευχαριστώ όμως που κατάφερες να απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Και πάλι νομίζω ότι έχεις καταλάβει ότι όλοι χαίρονται πάρα πολύ που σε βλέπουν και πάλι εδώ. Και ελπίζουμε ότι θα σε ξαναδούμε σύντομα. Brian, all the best. Okay, Ολοκληρώνεται τώρα η συνεδρία και κυκλισμένο των θυρών θα γίνει συνεδρία στο συντονιστό.